Bonjour mesdames et messieurs, je vous demande bien vouloir prendre place. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να καθίσετε και να συνεχίσετε τις συζητήσεις σας εκτός εθούσης και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή με την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Θέλω να σας πω ότι στα πλαίσια των ανταλλαγών απόψεων για την κρίση στο ΣΑΕΛ ε, θα συναντήσουμε όχι μόνο τους ε, εκπροσώπους της Γενικής Διευθύνσεως ΕΚΟ αλλά και άλλους που θα μας παρουσιάσουν τις θέσεις τους και τις αξιολογήσεις σχετικά με διάφορα θέματα όπως η διατροφή, ε, η κατάσταση των νέων κτλ. Ε, έχουμε λοιπόν μία γενική θεώρηση ε, ε, για την για την το θέμα της ανάπτυξης και επιπλέον θα έχουμε ε, διάφορες παρουσιάσεις ε, σχετικά με τα θέματα του ασύλου. Αν δεν έχετε ε, κάποια αντίρρηση θεωρούμε ότι ενεκρίθη η μερίσια διάταξη και έχετε και τα πρακτικά της συναντήσεως της 27 Μαΐου 2012. Ε, αν έχετε παρατηρήσεις ενημερώστε την ε, γραμματεία πριν τελειώσει η σημερινή συνεδρίαση διότι στη συνέχεια θα θεωρηθεί ότι έχει υιοθετηθεί και το πρακτικό. Επίσης έχετε τις συστάσεις και τις αποφάσεις που λήφθησαν στην ε, ε, συνάντηση της 27ης Μαρτίου. Αν έχετε παρατηρήσεις ενημερώστε τη γραμματεία πριν από το πέρας της σημερινής συνεδριάσεως διότι διαφορετικά θα θεωρηθούν ως ε, εγκριθέντα και τα θέματα αυτά. Λάβαμε μία ερώτηση από τον κύριο Φρανκ Μανέκ ε, σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Μανέκ δεν είναι εδώ, οπότε το ερώτημά του δεν θα συζητηθεί τώρα. Μετά, περνάμε στην παρουσίαση. Η κυρία Γκρέζ έλαβε τα έγγραφά της, εάν ναι, η κυρία Γκρέζ θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης ε, σχετικά με την εισήγηση έμβη για τις περιβαλλοντολογικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρισης σκισολιθικού αερίου και πετρελαίου και δίνω το λόγο στην κυρία Γκρέζ. Καλημέρα. Καλημέρα όλους. Ξέρω ότι είναι δύσκολη ζωή μία Δευτέρα απόγευμα. Θα μιλήσω γαλλικά. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι ένα σύνηθες θέμα προς εξέταση για μένα, διότι για τα θέματα των σχιστο ολυθικών αερίων ε, έχουμε ορισμένες προδιαγραφές αλλά ιδίως ε, στη χώρα μου τη Γαλλία υπάρχει μία ομόφωνη αντίρρηση όλης της πολιτικής τάξεως όλων των ερετών ε, είτε πρόκειται για δεξιά είτε για αριστερά παράταξη σχετικά με την εκμετάλλευση των σχιστολιθικών αερίων τόσο ανησυχούν για το θέμα αυτό. Εδώ όμως είμαστε στην Επιτροπή Ανάπτυξης και θέλω να τονίσω ότι το θέμα του σχιστολιθικού αερίου αναφέρεται πέραν ε, των συνόρων μας και είναι πολύ πιο ανησυχητική στις υποανάπτυξη χώρες για διάφορους λόγους. Καταρχήν γιατί δεν υπάρχει ίδια πρόσβαση στην ενημέρωση όπως έχουμε στη Γαλλία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και ιδίως διότι θα πληρώσουν ένα ακόμη πιο σοβαρό τίμημα και η εμπορική πολιτική τους τους υποκινεί για να μην καταρτήσουν μια πραγματική πλαισίωση οικολογική ε, των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στις χώρες τους. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία πρέπει να καταρτήσει ένα ρυθμιστικό υποχρεωτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες εξασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες. Δεν θα επεκταθώ τώρα στα παραδείγματα τα οποία συναντούμε, αλλά υπάρχουν ατυχή παραδείγματα σχετικά με την ε, εκμετάλλευση του πετρελαίου στις υποανάπτυξη χώρες και μπορώ να αναφέρω την ε, Αργεντινή για την κοιλάδα του Νιοκέν και τη Γουατεμάλα με την περιοχή του Πετέν ή μία σειρά από άλλα παραδείγματα όπου οι επιπτώσεις της ε, ε, εκμεταλλεύσεως του ορυκτού πλήτου ε, έχουν καταστρέψει και την βιοπικιλότητα και τις τοπικές συνθήκες. Άρα πρέπει να αποφεύγονται τέτοια παραδείγματα. Αλλά για το σχιστολιθικό αέριο πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση είναι χειρότερη και από την εκμετάλλευση του πετρελαίου διότι θα έχετε παρακολουθήσει την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον, για την υγεία και η εμπειρία των ε, Ηνωμένων Πολιτειών οδήγησε τον Απρίλιο του 2010 να, ε, ε, η πόλη της Νέας Υόρκη να σταματήσει τέτοιες δραστηριότητες και το ίδιο έχει ισχύσει και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, που δεν είναι λόγο δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε ή να στηρίξουμε μία δραστηριότητα η οποία κατά βάση είναι με την υλοποίηση του εβδόμου στόχου για την ανάπτυξη που είναι η διατήρηση του περιβάλλοντος για τις υποανάπτυξη χώρες καταρχήν θα πρόκειται για ένα σοβαρό κίνδυνο για την πρόσβαση στο νερό και υπενθυμίζω για όσους το αγνοούν πώς γίνεται η εξόριξη του σχιστολιθικού αερίου μέσω της του υδραυλικού κατακαιρματισμού όπου εμφυσούμε στο βάθος, στο υπέδαφος τόνους νερό δηλαδή τεράστιους πόρους υδάτινους και χημικά προϊόντα με μαζική έγχυση που καταστρέφουν τα πάντα. Σε εμά είναι δραματικό αλλά ακόμη χειρότερα στις υποανάπτυξη χώρες όπου αμφισβητείται η πρόσβαση στο νερό και επιπλέον στις υποανάπτυξη χώρες βλέπουμε ότι εδώ και λίγο χρόνο ήδη ε, υπάρχει ε, μία δέσμευση ε, των περιοχών για να υπάρξει εκμετάλλευση πράγμα που είναι εις βάρος και των ηθαγενών πληθυσμών και των φτωχών γεωργών. Πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν εμπεριέχει κάποιο εχέγγυο για τη διατήρηση και προστασία της ανθρώπινης υγείας και το περιβάλλον σχετικά με την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου. Γι' αυτό και είναι κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ ε, ε, βλέποντας την κατάσταση των υποανάπτυξη χωρών είμαστε υπεύθυνοι και θα πρέπει να επηρεάσουμε τις επιχειρήσεις μας για να χρησιμοποιήσουν πιο βιώσιμες μεθόδους και δεν φτάνει απλώς να αναφέρουμε εθελοντικές αρχές. Ε, ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποιο τρόπο πρόκειται να επιζητήσει και να βρει νέες ε, εναλλακτικές λύσεις για να εξασφαλίσει τα κοινωνικά δικαιώματα και τα περιβαλλοντολογικά δικαιώματα ε, όταν υπάρχει γενικός εκμετάλλευση πρώτων υλών και ιδιαιτέρως σχιστολιθικού αερίου. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή εν ονόματι της Επιτροπής Περιβάλλοντος και του ζητώ να λάβει υπόψη του τα σχόλιά μου και να τα ενσωματώ στην έκθεσή του. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε αν λίγο με συνέπαρε αυτό το θέμα αλλά πρέπει να υπολογίσουμε όταν μιλάμε για συστολιθικό αέριο στις υποανάπτυξη χώρες ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι ε, μία άνευ ε, εξέλιξη. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Νομίζω το θέμα αυτό είναι σοβαρό και άρα δεν υπάρχει λόγος να ζητάτε συγγνώμη. Και τώρα δίνω το λόγο σε όσους ε, θέλουν ε, να λάβουν το λόγο και ξεκινώ με τον κύριο Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκρές για τις ε, προτάσεις της σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και να πω ότι συμφωνώ με τα μέλη της Επιτροπής για κάποια από τα θέματα που και εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά όπως τα θεωρεί σημαντικά και η κυρία Γκρέσ η μορφή αυτή ενέργειας ε, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και είπα είναι η μόνη μέχρι στιγμής χώρα που χρησιμοποιεί αυτού του είδους την ενέργεια και υπάρχει ενδιαφέρον για την ε, Ασία, παραδείγματο χάρη ε, για το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί και εκεί, αλλά δεν έχει κάτι ξεκινήσει. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και την νομοθεσία εδώ. Είναι λίγο πρώιμο να πούμε αν χρειάζεται νέα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχουν υπάρχουν ε, πάρα πολλοί πραγματικοί κίνδυνοι ε, που αφορούν το περιβάλλον, ε, γιατί αυτή η μεθοδολογία, η τεχνική της υδρορογμάτωσης που χρησιμοποιείται είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, ιδίω γιατί καταναλώνεται πολύ μεγάλη ποσότητα νερού σε χώρε που πλήττονται από την ξηρασία, περιοχέ που πλήττονται από ξηρασία. Αυτό θα σχεράνει την κατάσταση. Εάν δεν ρυθμιστεί επίση μέθοδο, μπορεί να υπάρξει μόλυνση ε, των ε, υπόγειων ε, υδάτων, αλλά μέχρι και σεισμοί ή άλλες τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν από αυτή την τεχνική. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει πάντοτε να τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό τώρα το σχιστολιθικό αέριο το οποίο στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Γκρέσε, από τη βενζίνη έχει πολύ περισσότερη έκκληση διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα, Ολοκληρώνοντας, θεωρώ ότι η αναπτυξιακή βοήθεια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, και οποιαδήποτε άλλη φορείς δεν θα πρέπει να δίνουν χρήματα για, την, για το σχιστολιθικό αέριο σε υποανάπτυξη χώρες. Η κυρία Μάλιστα, το Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Είναι δύσκολο, κατά την άποψή μου, να μην συμμεριστεί κανείς ορισμένες από τις ανησυχίες σας. Και πράγματι υπάρχουν αρκετές ε, αποδείξεις για το ότι η εκμετάλλευση του σχεστολιφικού αερίου ε, λόγω των χημικών που χρησιμοποιούνται μπορεί να προκαλέσει και ε, την ε, ρήπανση των υδάτων, των υπόγειων, αλλά και την ατμοσφαιρική ρήπανση λόγω έκκλησης μεθανίου. Φαίνεται ότι Όλα αυτά γίνονται διότι το ίδιο το φρεάτιο δεν είναι απολύτως στεγανό. Δηλαδή υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που κλείονται από το ίδιο το πέτρο που περιέχει το αέριο. Αλλά και από τις εξορίξεις, στις εξορίξεις κάποιες φορές ε, δημιουργούνται ρήγματα και από αυτά τα ρήγματα περνούν οι χημικές ουσίες ε, και ρηπαίνουν τα υπόγεια ύδατα και διαφεύγει και το αέριο. Ε, ένα άλλο σχετικό αέριο είναι ότι αυτή η διαδικασία του fracking, της υδρορογμάτωσης δηλαδή, δημιουργεί πράγματι, μπορεί να προκαλέσει ε, σεισμούς. Και εμένα με ανησυχεί. Και μάλιστα η θέση της δικής μας κυβέρνησης, λαμβάνοντα υπόψη ότι όπου έγινε χρήση της τεχνικής αυτής της υδρορογμάτωσης, υπήρξαν σεισμικές δονήσεις στην περιοχή και φυσικά προκαλείται ανησυχία του πληθυσμού. Μπορεί να είναι μικρή ε, ε, κλίμακα, αλλά υπάρχουν θέματα οι σεισμοί, αλλά υπάρχουν θέματα για την αξιοπιστία αυτή τη μεθόδου. Τώρα, τούτου λεχθέντο, νομίζω ότι εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξετάζει η έκθεση αυτό. Έχουμε πολλά νομοθετήματα που στόχο έχουν να προστατεύσουν την ποιότητα των υδάτων και του αέρα. Και έχουμε λοιπόν η ολόκληρη δέσμη νομοθεσίας, νομοθετημάτων. Τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρούν όλη αυτή την νομοθεσία. Εάν και μάλιστα θα πρέπει να τηρήσουν και τις διατάξεις που σχετίζονται και με την εκμετάλλευση του και στο εφόσον να θελήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τι γίνεται όμως με τις τρίτες χώρες. Όλα αυτά τα νομοθετήματα τα οποία βάζουν περιορισμούς στην ε, εκμετάλλευση χιστολιθικού αερίου στην Ένωση δεν ισχύουν για τρίτε χώρες και θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να υπάρχει έλεγχος και να μην υπάρχει, αν θέλετε, μια αρπακτική καταχρηστική εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου που θα προκαλούσε καταστροφικές περιβαλλοντικές ε, ζημίες. Κάποιοι κάποιες τοποθεσίες όπως η Νότια Αφρική για τι οποίε προτείνεται η χρήση αυτή τη τεχνική, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λειψιδρία. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού για αυτή την ε, εξορρυκτική διαδικασία. Υπάρχει ανταγωνισμός και επίσης οι αγρότες, ο ντόπιο πληθυσμό ε, ε, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν πρόβλημα επάρκεια σε νερό αν χρησιμοποιηθεί και αυτή η τεχνική Επίσης αλήθεια είναι ότι και το αποτύπωμα ε, της ε, ε, του σχιστολιθικού αερίου στο περιβάλλον είναι πολύ μεγάλο, διότι αυτά τα φρεάτια, αυτές οι εξορίξεις δεν ε, διατηρούν για πολύ καιρό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να έχεις για πολλά χρόνια με ασφάλεια. Ουσιαστικά πρέπει να προχωρήσει όλο και περισσότερο, γιατί εξαντλείται το αέριο στο πέτρωμα, πρέπει να προχωράσει σε μεγαλύτερο βάθο και άρα αυξάνονται και, ε, αυξάνεται και το μέγεθος της καταστροφής που, που προκαλείται με αυτή τη μέθοδο. Και ε, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να, να βαθμιστεί το περιβάλλον για να προστατευτεί η βιοπικιλότητα. Όλα αυτά είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Ιδίω ό,τι αφορά την εκμετάλλευση σε τρίτες χώρες. Και ένα πιο γενικό σχόλιο τι επιπτώσει μπορεί να έχει όλη αυτή η διαδικασία για την αλλαγή του κλίματος. Αυτό με ανησυχεί. Λόγω της μεθόδου ε, της παραγωγής και του αερίου από το σχιστόλιθο, έχει μάλλον και με σοβαρότερο, μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με πιο συμβατικές ε, πηγές. Λόγω των χημικών ε, ουσιών και της ενέργειας που απαιτείται για την εξόριξη του αερίου. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αμμώδεις πίσες. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά εκλείονται στην ατμόσφαιρα και τελικά είναι ορυκτό καύσιμο το αέριο. Και παρότι μπορεί να εκλείεται μικρότερη ποσότητα ε, του άνθρακα από αυτό όταν το καίουμε σε σχέση με τον άνθρακα, αλλά μέχρι το 2050 εμείς θέλουμε να μειώσουμε ή τέλος πάντων να καταργήσουμε τη χρήση ε, του άνθρακα. Και δεν νομίζω ότι αυτή είναι η βέλτιστη λύση μακροπρόθεσμα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες καταστροφές. Πρέπει να το προσέξουμε λοιπόν. Και αυτό που με ανησυχεί κυρίως είναι πώς ε, ε, και γιατί μπορεί, μάλλον πώς μπορούμε να κάνουμε υπεύθυνα χρήση αυτής της τεχνολογίας μέσω της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο μέσο. Θα μιλήσω εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι ουδέτερη σε σχέση με την εκμετάλλευση αυτής της μεθόδου φυσικού αερίου έχουμε ε, μετά από εξέταση των διαθέσιμων πληροφοριών ότι η υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται και στην περίπτωση ανείχνευσης μη συμβατικών τρόπων εξαγωγής αερίου, μεταξύ των οποίων και ε, του φυσικού αερίου από σχιστολιθικούς τόπους. Λόγω όμως των περιορισμένων γνώσεων που έχουμε σχετικά με τις τεχνολογίες αυτές που βρίσκονται στην αρχή της ανάπτυξής τους, τουλάχιστον στην Ευρώπη, θα ήταν προώρο να πούμε αν το υπάρχον κοινοτικό πλαίσιο διασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έδωσε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για το νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται στα προγράμματα αυτά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει περαιτέρω μελέτες για να αξιολογήσει πιθανούς κινδύνους σχετικά με τις πρακτικές αυτές. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη και θα συνεχίσει και τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκομένους και όπου χρειάζεται θα δώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμέ που απαιτούνται. Ε, περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις δραστηριότητες και τις συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά και στη δική σας Επιτροπή. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρέζα έχει ξανά το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Είδα ποια σημεία χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης η σεισμολογική κίνδυνη σαν παράδειγμα, οι συνέπειες στο τοπίο, στην εικόνα του φυσικού χώρου. Και εγώ έχω ταξιδέψει τα τελευταία δέκα χρόνια στο Wyoming επανειλημμένα. Όταν βλέπω κάποια τοπία σήμερα δεν αναγνωρίζω τίποτα. Ε, δεν ξέρω τι δυνατότητα υπάρχει αποκατάσταση των χώρων, να πολύ αμφιβάλλω. Και τέλος να πω στον σοσιαλιστή συνάδελφο, ο οποίος έχει επιμείνει στις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών και στο θέμα το πολύ αρνητικό δυστυχώς και για την εκπομπή αερίων και αυτό ισχύει και για τις ασφαλτούχες άμμος. Σχετικά τώρα με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιμένω ακόμα το αποτέλεσμα των μελετών που αυτή τη στιγμή διεξάγονται. Δεν σας κρύβω ότι η δική μου θέση είναι ότι χρειαζόμαστε μια νομοθεσία η οποία να είναι πιο σαφής γύρω από τη σχιστολιθικά αέρια. Ε, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ε, και νομικά πλαίσια όπως και η συνθήκη ότι προβλέπει το Natura 2000 κτλ. Αλλά οι επιχειρήσεις μας θα μπορούσαν να μην σεβαστούν τέτοιου είδους οδηγίες όταν εγκαθίστανται σε υποανάπτυξη χώρες. Και σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο ακόμα και στην ίδια την Ευρώπη να πλαισιώσουμε με ακριβέστερο τρόπο το θέμα της εξαγωγής αερίου από σχιστόρυθο. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερώτηση για την οποία δεν πήρα απάντηση για τις υποανάπτυξη χώρες. Γνωρίζουμε ότι στις υποανάπτυξη χώρες, είχα πάει στο Σαχέλ πρόσφατα, ο κόσμος πεθαίνει λόγω λειψιδρίας. Συνεπώς λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να ψάχνουμε για αέριο σε αυτές τις περιοχές. Έχετε μια απάντηση να μας δώσετε γύρω από αυτό γιατί είναι εντελώς διαφορετική εκεί η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω απάντηση για το ερώτημά σας δυστυχώς. Ε, αυτό είναι η απάντηση την οποία επιζητούσα. Ο κύριος Βάγκελ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να μην ε, χρησιμοποιεί τον όρο ότι είμαστε ε, ουδέτεροι. Εάν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα δεν μπορούμε να παραμένουμε ουδέτεροι όταν γνωρίζετε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρόκειται να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες στις ε, εμπλεκόμενες χώρες και στις φτωχότερες χώρες, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα έπρεπε να έχει μία πιο επικοδομητική αντιμετώπιση των θέματων αυτών και να μην παραμένει ουδέτερη. Ευχαριστώ και καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί το θέμα αυτό, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, οξίες ε, και ε, πολύ σημαντικές. Οπότε η, αύριο τελειώνει η προθεσμία ε, στις 8 Μαΐου το μεσημέρι. Τώρα αναφερόμαστε σε συνδυασμό επιχορηγήσεων με δάνεια για την εξωτερική συνεργασία για την ανάπτυξη. Θα υπάρξει μία παρουσίαση του θέματος από την ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν τέλειωσα όμως και σιωπώ διότι εδώ βλέπω και υπάρχουν πολλά ε, συζητήσεις και δεν ξέρω ε, εγώ εάν θέλω να πω κάτι εις ε, τη γραμματέα ψιθυρίζω δεν μιλάω δυνατά λοιπόν Συνδυασμό επιχορηγήσεων με δάνεια για την εξωτερική συνεργασία και την ανάπτυξη. Ξεκινάμε το θέμα αυτό με μία παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βάγκε Πλάνας Επιτροπής και την ε, κυρία Τζάκι Τζαν οι οποίοι ήρθαν να κάνουν την παρουσίασή τους σχετικά με τις περιφερειακές δυνατότητες συνδυασμού επιχορηγήσεων με δάνεια. Έχετε 15-20 λεφτά στη σειρά την οποία επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Αν με επιτρέπετε θα μιλήσω αγγλικά, κυρία Πρόεδρε, γιατί σε αυτή τη γλώσσα έχουμε προετοιμάσει την παρουσίασή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι αυτά τα οποία θα σας παρουσιάσω αποτελούν λίγο πολύ τα, το περιεχόμενο ενός κειμένου το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε. Ακούσαμε για κάποιους μηχανισμούς συνδυασμού και κατά το παρελθόν και δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα το συζητήσουμε. Φαντάζομαι ότι και στο άμεσο μέλλον θα χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα επικεντρωθούμε στα βασικά αυτού του συνδυασμού επιχορηγήσεων για να μην ε, ξεπεράσουμε και το χρόνο που μας έχετε διαθέσει. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι βασικές στοιχείες των συνδυασμών. Γιατί ένα μεγάλο μέρος αναπτυξικής συνεργασίας ε, το μεταφέρουμε στους μηχανισμούς συνδυασμού. Για να σας δώσουμε κάποιες βασικές ιδέες, αλλά και τους βασικούς ε, στόχους, έχουμε προετοιμάσει κάποιες διαφάνειες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες μαζικές ε, εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η φτώχεια. Και το λιγότερο που μπορεί να πει κανεί είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, πολύ μεγάλους περιορισμούς για τα δημόσια κονδύλια τα οποία δίνονται στην αναπτυξιακή συνεργασία. Κονδύλια τα οποία τουλάχιστον ε, δεν αυξάνονται στην ταχύτητα που θα θέλαμε, αν, δεν αυξα... αν αυξάνονται και καθόλου. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το συνδυασμό για να έχουμε ένα αποτέλεσμα μόχλευσης. Δεν προσπαθούμε να πετύχουμε με τις επιχορηγήσεις μας προσπαθούμε να ε, έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μέσω μόχλευσης για να μην χρειαστούν πρόσθετοι πόροι είτε από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς ε, οργανισμούς. Η χρήση των επιχορηγήσεων μπορεί να κάνει πιο βιώσιμα κάποια σχέδια. Ουσιαστικά αυτή οι επιδοτήσεις είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ Θα μπορούσε κανείς να πει, έτσι για να ε, μην μακρηγορώ, ότι ο συνδυασμός ουσιαστικά σημαίνει επιχορηγήσεις συν δάνεια ή πιστώσεις. Δηλαδή έχουμε κονδύλια για επιχορηγήσεις και τα συνδυάζουμε με πιστώσεις, ε, με δάνεια είτε από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς είτε από άλλους δωρητές, από άλλους χρηματοδότες. Εν γέννη, ε, με τους χρηματοοικονομικούς πόρους που έχουμε να κάνουμε και θα το δείτε αργότερα σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ε, εκεί μπορεί να έχουμε κάποια, ε, κάποιες διαφορές. Έχουμε πάντως χρήση κοινοτικών πόρων και αυτή είναι η απαρχή ε, του συνδυασμού, αλλά αυτοί οι πόροι μπορούν να συνδυαστούν με επιχορηγήσεις από άλλους χρηματοδότες και κανονικά Έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Ίδρυμα, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη της ε, χρηματοδότησης του σχεδίου ή σε κάποιες περιπτώσεις μη ευρωπαϊκά δημόσια οικονομικά ιδρύματα όπως παραδείγματος χάρη τράπεζες ε, περιφερειακής ανάπτυξης στις διάφορες περιοχές όπου εργαζόμαστε. Ή σε κάποιες περιοχές μπορεί να υπάρχουν εμπορικοί επενδυτές ή επενδυτές ή ιδιωτικές ε, εμπορικές τράπεζες. Ή οι πόροι μπορεί να αυξηθούν με ίδιους πόρους των δικαιούχων χωρών. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι αυτοί οι πόροι περιλαμβάνονται, αλλά πάντα θα υπάρχει ένα συνδυασμός ορισμένων από αυτά τα στοιχεία. Και θα πρέπει να έχετε υπόψη σα ότι ο μηχανισμός συνδυασμού είναι ένας μηχανισμός συνδυασμού, επαναλαμβάνω, που έχουμε ένα σκέλος επιχορήγηση και ένα σκέλος δάνειο ή πίστοση. Ποιοι είναι οι στόχοι της ε, πρακτικής αυτής. Πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, ο στόχος μας είναι να έχουμε μια χρηματοοικονομική μόχλευση, να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις επιχορηγήσεις μας για να ε, μοχλεύσουμε περισσότερους ε, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για να έχουμε μεγαλύτερο αναπτυξιακό αντίκτυπο. Να πολλαπλασιάσουμε δηλαδή το οικονομικό αποτέλεσμα των επιχορηγήσεων. Θέλουμε να έχουμε πρόσθετα κονδύλια, τα οποία θα προσθέσουμε στις επιχορηγήσεις μας. Πέραν τούτου, μπορεί να έχουμε και μη χρηματοοικονομική μόχλευση. Δηλαδή, παρέχοντας ε, κονδύλια μέσω του μηχανισμού συνδυασμού βελτιώνουμε είτε την ταχύτητα είτε τη βιωσιμότητα ενός σχεδίου. Παραδείγματο χάρη παρέχοντας τεχνική βοήθεια η οποία επιταχύνει την ε, προπαρασκευή του σχεδίου ή το βελτιώνει. Μια άλλη δυνατότητα είναι μεγαλύτερη οικονομική πειθαρχία και ιδιοκτησία. Δηλαδή ότι οι μηχανισμοί ε, το ότι οι μηχανισμοί συνδυασμού περιλαμβάνουν και το στοιχείο της πίστη, της πίστοσης πάντοτε, αυτό ε, αναγκάζει την δικαιούχο χώρα να σκεφτεί το πώς θα επιστρέψει ε, τα χρήματα αυτά. Και έχει μεγαλύτερη λοιπόν βιοκτησία και περισσότερο αυτό το, σχέδιο. Το γεγονός επίσης ότι συσχετίζουμε με ε, επιδοτήσεις από την κοινότητα, τους πόρους αυτούς, αυτό βοηθά να ε, υποστηριχθούν και οι μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό κυρίως όταν εξασφαλίζουμε το ότι η φιλοσοφία όλων αυτών των μηχανισμών συμφωνούν συμφωνεί με τους στόχους ε, της ε, κοινωτικής αναπτυξιακής πολιτικής. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ένας δεύτερος στόχος του συνδυασμού, αν θέλετε καλύτερα, το δεύτερο αποτέλεσμα του συνδυασμού είναι ότι προωθεί τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων και φορέων που εργάζονται στο αναπτυξιακό πεδίο. Αυτό συμβαίνει σίγουρα μεταξύ Ευρωπαίων και μη Ευρωπαίων παραγόντων, εταίρων δηλαδή όπως είναι τράπεζες που δεν είναι ευρωπαϊκές, αλλά κάτι σημαντικό επίσης δημιουργεί και ένα σύνδεσμο μεταξύ των χρηματοδοτών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Διότι αρχικά πρόκειται και δύο ξεχωριστού κόσμου. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια όλο και περισσότερο αυξάνεται ο συντονισμό με αυτού ε, του ε, δωρητέ που παρέχουν δηλαδή επιδοτήσει, επιχορηγήσει και αυτού που παρέχουν δάνεια ή πιστώσει. τέλο. και με το μέγεθο των σχεδίων, γιατί μιλάμε για σχέδια υποδομών. Με το μέγεθο λοιπόν σίγουρα αυξάνεται η προβολή των σχεδίων και η ευρωπαϊκή του διάσταση. Αυτό το γράφημα είναι αρκετά τεχνικό και δεν θέλω να μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, αλλά να τονίσω ότι από την ταυτοποίηση μέχρι την αξιολόγηση ενό οδήποτε σχεδίου. Η Κομισιόν ελέγχει όλα τα στάδια με κάποιες μικρές διαφορές από ό,τι κάνουμε για τις επιδοτήσεις. Έχουμε ένα στάδιο της υλοποίηση αυτών των συνδυασμένων σχεδίων, το οποίο μπορεί να εκχωρηθεί, να ανατεθεί ε, σε έναν ε, χρηματοδοτικό οργανισμό. Αν θέλουμε όμως να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειάς μας, κάνουμε εξολογήσεις εκ των προτέρων, σε ό,τι αφορά την ικανότητα, τη λογιστική κτλ. Και μόνο πιστοποιημένοι χρηματοδοτικοί, ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτού του εξάντε ελέγχους και εξολογήσεις. Κάτι άλλο που θέλουμε είναι να συμμετέχουν που θα έπρεπε ούτω ή άλλω, όλο και περισσότερε αντιπροσωπείς τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη τη διαδικασία τη διαπραγματεύση με του τρίτου χώρε, την προετοιμασία του σχεδίου, αρχίζοντα βέβαια με την ταυτοποίηση και καταλήγοντα και στην ε, συνέχεια που δίνεται στην ε, υλοποίηση, στην παρακολούθηση. Το χρηματοπιστωτικό έδρυμα παίζει ρόλο γιατί ουσιαστικά υλοποιεί αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και ε, αυτά διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Θα επανέλθω αργότερα σε αυτά τα σημεία, γιατί ίσως είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσετε τη διαφάνεια αυτή. Και έρχομαι σε ένα άλλο slide για να σας πω ότι όταν λαμβάνουμε ένα σχέδιο προς χρηματοδότηση και αν πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά, κάνουμε κάποιους ελέγχους όλο και περισσότερο αυξάνουμε τη διαδικασία του screening, της διαλογής δηλαδή των έργων που μας υποβάλλονται. Πρώτα απ' όλα, τα έργα αυτά πρέπει να συμφωνούμε με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Πολιτικής. Επίσης, θα πρέπει τα έργα να πληρούν ε, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που έχουμε θεσπίσει και κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να αιτιολογείται επαρκώ η ανάγκη για τη χρήση των ε, επιχορηγήσεων. Αυτό είναι ιδίως ε, σημαντικό εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσει τη αγορά μέσω της παροχής ε, επιχορήγηση σε συνδυασμό με ένα δάνειο μια πίστοση. Να σα πω ότι όλο και πιο πολύ αντιλαμβανόμαστε το γεγονό ότι τα ζητήματα χρέου πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν το επαναλαμβάνω, εμείς παρέχουμε χρηματοδότηση υπομορφή επιχορήγηση που συνδυάζεται με δάνεια ή πίστοση, άρα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και αυτό το ζήτημα το αντιμετωπίζουμε με όλο και μεγαλύτερη σοβαρότητα. Τώρα, πώς ε, γίνεται η υποβολή των σχεδίων ε, στους περιφερειακούς ε, φορείς. Ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα είναι αυτό που πάντοτε υποβάλλει τα έργα. Και έχουμε την έννοια του lead financier. Αυτό είναι ένα ίδρυμα σημαντικό χρηματοπιστωτικό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι ο βασικός μας εταίρος, η BERD, η Τράπεζα για την Συγκρότηση και την Ανάπτυξη, ή εθνικοί οργανισμοί, αναπτυξιακοί οργανισμοί το KFW, Sims και τα λοιπά. Βλέπετε και τις ε, αντίστοιχες εθνικές ε, οντότητες. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης, περιφερειακές ε, τράπεζες ανάπτυξης μπορεί και αυτές να είναι πλήρω μέλη αυτού του μηχανισμού, όπως είναι η, τράπεζα, η Αφρικανική Τράπεζα για την Ανάπτυξη και άλλες. Και το ίδιο θα γίνει με την Καραϊβική, με την Διαμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα ότι θα εγκρίνουμε ένα μηχανισμό για την καραϊβική όπου να είναι. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι παρατηρητές. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να παρουσιάζουν ως lead financiers, ε, ως ε, βασική δηλαδή στο πρόγραμμα, αλλά συμμετέχουν. Όπως η Διαμερικανική Αναπτυξική Τράπεζα και η Κεντρική Αμερικανική Τράπεζα για την Οικονομική Ολοκλήρωση, Corporación Andina de Fomento για τη Λατινική Αμερική κτλ. Να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι εν γέννη έχουμε ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο παρουσιάζει το έργο και ζητά επιχορήγηση η οποία θα προσθεθεί στη χρηματοδότηση του σχεδίου. Πολλές φορές όμως δεν είναι μόνο αυτό το βασικό χρηματοδοτικό ίδρυμα που συμμετέχει, μπορεί να υπάρχουν, όπως είπα, περιφερειακές τράπεζες ή εμπορικές τράπεζες ή, άλλου είδους χρηματοδότηση. Τρία, ε, τρεις πυλώνες έχει η καρτική δομή, η δομή διακυβέρνησης. Πρώτα απ' όλα, έχουμε έγκριση ενός προγράμματος για μια συγκεκριμένη περιοχή και έπειτα κάθε πρόγραμμα, κάθε έργο το οποίο υποβάλλεται σε αυτούς τους περιφερειακούς μηχανισμούς, στα regional facilities, περνάει από μια διπλή ανάλυση. Η πρώτη ανάλυση είναι, ε, γίνεται από ένα τεχνικό φορέα. Finance Intermediary Group, τέλο πάντων είναι μια ενδιάμεση ομάδα, δεν έχει το σημασία το όνομα που έχει, αλλά κυρίως ότι πρόκειται για ένα τεχνικό φορέα που αναλύει τεχνικά το έργο. Βλέπει δηλαδή και τα οικονομικά στοιχεία αλλά και τα αναπτυξιακά στοιχεία του έργου. Με την Επιτροπή να προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού του φορέα. Αν θεωρούμε ότι είναι αρκετά όριμα τα έργα, τα υποβάλλουμε σε ένα δεύτερο φορέα, στο Συμβούλιο Board, που συνήθως δίνει το πράσινο φως ή το κόκκινο φως, ανάλογα βέβαια με τα με την άποψη των κρατών μελών. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρετε ότι έχουμε δύο στρώματα. Το πρώτο είναι τεχνικό, όπου εκπροσωπούνται οι τράπεζε και την Προεδρία έχει η Κομισιόν και αντιπρόεδρο είναι η ΕΕΠ, ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έπειτα δεύτερο στρώμα το Συμβούλιο, όπου τα κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται λαμβάνουν την απόφαση για το κατά πόσον θα πρέπει να δοθεί η ε, επιχορήγηση στο ε, προκείμενο έργο. Επίσης, μπορεί το Συμβούλιο να συνέλθει, να συνεδριάσει και για στρατηγικούς σκοπούς. Υπάρχει στο πλαίσιο του μηχανισμού ένα έγγραφο στρατηγικού προσανατολισμού που αναφέρει ποιοι είναι οι τομεί όπου θέλουμε να εργαστούμε, ποιε είναι οι βασικές προτεραιότητες για την περιοχή. πώ θα εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά συνάδουν με του περιφερειακούς στόχου κτλ. Όλα αυτά γίνονται σε συνδυασμό με τι δικαιούχου χώρε και με τα κράτη-μέλη. Mm. και σε αιτήσια βάση γίνεται η ανάλυση για να δούμε κατά πόσον ε, ισχύουν ή όχι οι στόχοι που έχουμε θέσει, αν πρέπει να αλλάξουν, να τροποποιηθούν, να προσθεθούν νέες προτεραιότητες κτλ. Το κομμάτι που ίσως να σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η γενική εικόνα, η ευρύτερη εικόνα. Τι γίνεται λοιπόν με αυτούς ε, τους ε, περιφερειακούς ε, συνδυασμούς, περιφερειακούς μηχανισμούς συνδυασμού επιχορηγήσεων με δάνειο. Με την έγκριση αυτών των νέων μηχανισμών για την Ασία, για την Καραϊβική, για τον Ειρηνικό, έχουμε καταφέρει πρακτικά να έχουμε μια παγκόσμια κάλυψη των επενδυτικών μηχανισμών Έχουμε και ένα άλλο Trust Fund ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, δημιουργήθηκε το 2007. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει την Προεδρία. Επίσης έχουμε τον επενδυτικό μηχανισμό γειτονίας που δημιουργήθηκε το 2008 και έπειτα το 2010 επενδυτικός μηχανισμός για την Κεντρική Ασία και Λατινοαμερικανικός επενδυτικός μηχανισμός. Εγκρίθηκαν εκείνη τη χρονιά λοιπόν και τα δύο αυτά μέσα. Και πρέπει να σας πω ότι η επιτυχία του μοντέλου έχει ως αποτέλεσμα κάποιες χώρες που είναι εκτός της εικόνας, εκτός του τοπίου αυτού, ζητούν ε, αντίστοιχα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη, που το παρόντο διαπραγματευόμαστε επενδυτικό πρόγραμμα εθνικού τύπου με την Νότια Αφρική. Έχουμε λάβει έτοιμα για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε με τα ίδια εργαλεία στην Τουρκία. Αυτά σας τα λέω για να αποκομίσετε μία εικόνα του πόσο επιτυχημένο αυτό το μονοπάτι, ε, αυτή η πορεία των ε, μηχανισμών που σας παρουσιάζουμε. Πόσα χρήματα πηγαίνουν σε, αυτό, σε αυτούς τους μηχανισμούς. Το Trust Fund υποδομών ομήρια ε, πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά περιλαμβάνει και τη συμμετοχή από τα κράτη-μέλη. 400 εκατομμύρια ευρώ είναι για το σχετικό με την Αφρική. Ε, για τον επενδυτικό μηχανισμό με την Ασία είναι καινούριο μηχανισμό και είναι 30 εκατομμύρια το ποσό για τα έτη έως το 2012 τα πρώτα χρόνια μικρό το ποσό. Το ΙΦΚΑ για την Κεντρική Ασία έχουμε 65 εκατομμύρια. Για τη Λατινική Αμερική ο επενδυτικός μηχανισμός είναι 125 εκατομμύρια και ίσως η καλύτερη πρικοδότηση, μεγαλύτερη πρικοδότηση είναι για τη γειτονία, για, το μέσο, για τον επενδυτικό ε, μηχανισμό, για τη γειτονία 740 εκατομμύρια και 70 από τα κράτη-μέλη μέσω της συμμετοχής τους. Νομίζω ότι αυτή η διαφάνεια είναι η πιο σημαντική. Εάν προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε το σύνολο των ποσών, το οποίο έχουμε δαπανίσει από το 2007, στις τέσσερις πρώτες, στα τέσσερα πρώτα μέσα, βλέπω ότι έχουμε εδώ 760 εκατομμύρια δάνεια Ε, συγγνώμη, αν βάλετε μαζί τις επιδοτήσεις, τα δάνεια και τα επενδυτικά μέσα, φτάνουμε περίπου σε 26 δις. Από τα 26 δις, τα 10 δίδουν ε, τα ανεξάρτητα πιστοτικά όργανα. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Εδώ είναι η μόχλευση στην οποία αναφέρθηκα. Μέσω των ε, επιδοτήσεων των κοινοτικών. Νομίζω ότι αυτό δείχνει την επιτυχία μέχρι τώρα, μέχρι τώρα επιμένω, των επενδυτικών μας μέσων στις τέσσερις περιφέρειες. Ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σας δείξω τους τομείς οι οποίοι καλύπτονται. Είναι παρόμοιοι σε όλα τα μέσα άνω του 30%, του τρίτου συγγνώμη πηγαίνει στις μεταφορές. Ένα τρίτο πηγαίνει επίσης και στον τομέα της αηφορίας και της ενέργειας. 16% στην εξυγίανση των υδάτινων πόρων. Ένα μικρό ποσό σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε στήριξη μικρομεσαίων και αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε αν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα ένα μικρό τμήμα επίσης στην πληροφορική και ένα επίσης μικρό κομμάτι στις κοινωνικές υποδομές. Συζήταγα σήμερα το πρωί με τον εισηγητή του DCI και εξήγησα τις δυσκολίες που έχουμε όταν μπορεί, προσπαθεί κανείς να πάρει δάνεια στον κοινωνικό τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στο μέλλον. Οι δυσκολίες εκεί είναι πολλές. Να πω επίσης όπως έχει πει και πει το έχει βάλει και τις, τα χαρακτηριστικά θα έλεγα για τον έλεγχο όλων των προγραμμάτων, όλων των μέσων σε σχέση με την επιρροή που έχουν ή δεν έχουν για τις κλιματολογικές αλλαγές. Το 60% των προγραμμάτων ανήκουν σε κατηγορίες οι οποίες επηρεάζουν θετικά την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Τώρα, ο τύπος των επιδοτήσεων, το 1 τρίτο πηγαίνει σε άμεσες επενδύσεις, χρηματοδοτούμε άμεσα τις δημόσιες επενδύσεις, 33% πηγαίνει σε τεχνική βοήθεια, είτε στην αρχή του προγράμματος αλλά και στην συνέχεια, στην εφαρμογή του προγράμματος μπορούμε να δώσουμε τεχνική βοήθεια. Το 1 τέταρτο πηγαίνει σε επιδότηση των επιτοκίων, μειώνουμε το κόστος των δανείων και ένα μικρό τμήμα πηγαίνει σε ρίσκ και κεφάλαια κινδύνου και σε εγγύησεις. Είναι κάτι που πρέπει να καλύψουμε αν θέλουμε να συνεργαστούμε και να επηρεάσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου, στην συνάδελφό μου, η οποία θα σας δώσει κάποια παραδείγματα. Είπα ότι αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε 100 προγράμματα τουλάχιστον. Ε, εδώ θα σας δώσουμε μόνο ένα μικρό, μικρό δείγμα αυτών τα οποία κάνουμε. Τζάκι, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μαζί με την Επιτροπή παρουσιάζουμε κάποια από τα προγράμματα Τα παραδείγματα που θα σας δώσω δίνουν τη σημασία θα έλεγα των μηχανισμών που χρησιμοποιούμε και η πρόσβαση σε επιδοτήσεις και μέσω της τράπεζας ή μέσω άλλων μέσων χρηματοδοτικών. Το θέμα είναι να προχωρήσουν τα προγράμματα αυτά. Αυτό έχει σημασία ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες όπου είναι οι παρεμβάσεις αυτές απαραίτητο για να καλυφθούν προβλήματα και να διασφαλίσουμε επίσης ότι τα προγράμματα είναι σωστά προπαρασκευασμένα. Απαιτείται να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά τα ε, χρηματοδοτικά μέσα και μεγαλύτερη διαφάνεια. Λοιπόν, τρία προγράμματα. Το πρώτο αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ένα ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη και στην Νότια Ευρώπη. Εδώ υπάρχει συνδυασμός ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χρησιμοποιούμε στα Δυτικά Βαλκάνια σαν παράδειγμα και το Ταμείο Γειτονίας, αυτό που λέμε έτσι, σαν ένα πρώτο στάδιο παρέμβασης. Αυτό είναι ένα σωστός τρόπος για να προσελκύσουμε και άλλους επενδυτές, λειτουργεί καταλητικά η χρήση αυτών των μέσων γιατί μειώνεται ο κίνδυνος. Η μόχλευση στην οποία προαναφερθήκαμε νομίζω έχει μεγάλη σημασία εδώ. Βλέπετε εδώ ότι φτάνουμε 70 εκατομμύρια συνολικά, 10 εκατομμύρια είναι επιδοτήσεις. Συνεργαζόμαστε και με επιστοτικούς οργανισμούς όπως η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Αυστρίας. Ένα άλλο θέμα είναι, είναι η μονάδα παραγωγής με χρήση του ηλίου στο Ουαρζαζάτ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μεγάλο βάρος, σημαντική εικόνα και υποστηρίζει τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας στο Μαρόκο. Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας και την αποφυγή εκπομπής καυσαερίων διοξίδιου άνθρακα. Είναι τμήμα του Μαροκινού Ηλιακού Προγράμματος. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό θα είναι το μεγαλύτερο και το ισχυρότερο στην Βόρεια Αφρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόγραμμα ωφελείται από μια άμεση επιδότηση το οποίο μειώνει το κόστος του ηλεκτρισμού και καθιστά οικονομικά ελκυστικό το πρόγραμμα. 30 εκατομμύρια έχει δώσει η Επιτροπή έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ για τα μέσα τα οποία συνδυάζουμε. Υπάρχει θα έλεγα ένα σύστημα αμοιβαία στήριξης. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τα ισχυρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση επιμέρους και έτσι προσπαθούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής μας. Το τελευταίο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρέμβασης στην Αφρική και εδώ συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με άλλα χρηματικά μέσα ευρωπαϊκά. Βοηθά την διασύνδεση ενέργειας στον τομέα της ενέργειας από τη Ζάμπια μέχρι την Αμίμπια καλύπτει τη συνεργασία και ε, σε ύψος 50 εκατομμυρίων ευρώ με την Υπηρεσία Ενέργειας της Ναμίμπια και με διεθνείς άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Να προσθέσω εδώ κάτι. I think that, um, the main... Οι βασικές ανησυχίες που έχουμε σε αυτή τη φάση είναι το πώς θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τη χρήση των υπαρχόντων μέσων μέσω ακριβώς καλύτερων μέσων συνεργασίας να ε, προσελκύσουμε περισσότερα αναπτυξιακά πιστοτικά ιδρύματα, να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις νέες μίξεις μέσων ε, και της χρήσης αυτών σε περιφερειακό επίπεδο, και επίσης να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση από πλευράς του ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά βρίσκονται υπό συζήτηση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη και συνεργασία που θα συναντηθεί πάρα πολύ σύντομα. Και αν καταλήξουμε στη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας, τότε αυτά τα θέματα, τα τεχνικά που αντιμετωπίζουμε θα τύχουν περαιτέρω εξέταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κι εγώ. Και Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέζε αν επιθυμεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη φορά δεν μιλώ για λογαριασμό μου, αλλά για τον συνάδελφο Μπατ Στες, ο οποίος είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα οικογενειακό και δεν μπόρεσε να έρθει και απλώς θα σας διαβάσω το έγγραφο το οποίο πρόκειτο να παρουσιάσει και το οποίο έχει επεξεργαστεί με τη γραμματεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήρτισε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως και των κρατών μελών για να αξιολογήσει το κόστος που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο μέχρι τα μέσα του 2012 για να υπάρξει μία ανάμιξη η οποία θα βελτιώσει τη συνεργασία και προβλέπουμε ότι θα υπάρχει υπάρχει μία βελτίωση της προβολής και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων οργανισμών που συμμετέχουν διότι ο καθένας θα προωθήσει την εξωτερική δράση σε σχέση με τους στόχους της πολιτικής και αυτό θα επιτευχθεί με την ε, συγκέντρωση των πόρων και ε, των εμπειριών των βασικών ε, εμπλεκομένων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και όσον αφορά την δομή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί μία επιτροπή η οποία θα οργανώσει συνεδριάσεις υψηλού επίπεδου για να καθοριστεί ο συγκεκριμένος ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εις ε, την προσπάθεια αυτή και ε, στη συνεργασία με τους δημοσιονομικούς οργανισμούς. Ένα άλλο θέμα ήταν η νομική ε, βάση της πλατφόρμας αυτής και θεώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν χρειάζεται ειδικό νομικό πλαίσιο, αλλά σημαντικές Σημαντικά επιχειρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι μέχρι στιγμής η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είχε προβλεφθεί και προβλέπεται απλώς ότι θα λαμβάνει μία ετήσια έκθεση για την εργασία της πλατφόρμας, πράγμα το οποίο της ομάδος δηλαδή, πράγμα το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτήματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα υπάρχει επαρκής ε, συναπόφαση και έλεγχος ε, του προϋπολογισμού και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο μείγμα αυτό. Πώς ε, θα εξασφαλιστούν τα δικαιώματα εφόσον πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν θα αφιερωθεί σε ένα αμυγός κοινοτικό χώρο. Επίσης πώς θα εξεταχθούν οι δυνατότητες να αναμειχθούν οι μηχανισμοί με μόχλευση σε διάφορους δύσκολους τομείς όπως είναι ε, ο κοινωνικός τομέας, οι βιώσιμες ενέργειες και ούτω καθεξής. Ε, πώς θα μπορέσει να προωθηθεί μία πρωτοβουλία σε ε, μία οικονομική οικονομικο-κοινωνική ε, επιφάνεια. Πώς ε, θα αξιολογήσουμε το αμίγμα πρέπει να υπάρχει ένα τυποποιημένο μήνυμα το οποίο ε, θα αξιολογεί τις λειτουργίες του μείγματος και θα περιλαμβάνει ποιοτικούς δείκτες και ε, θα προβλέπει και κοινωνικές προόδους. Ε, θα, πρέπει να γίνει μία μελέτη των επιπτώσεων για τη συνεργασία με τον ειδικό τομέα, να υπάρχει μία διευκρίνηση και ιδίω όσον αφορά τη συμμετοχή του ειδικοτικού τομέα η οποία έχει αναφερθεί ως ε, ο χώρος OECD-DSE από τους ειδικού. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να παρέμβει. Όχι. Μήπως θέλει η Επιτροπή να απαντήσει στο σχόλιο το οποίο έγινε. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις. Νομίζω ότι ο στόχος της παρουσίας μας σήμερα είναι να παρουσιάσουμε μια, μια ε, γενική παρουσίαση ε, το, ε, της συνεργασίας. Η Επιτροπή Ανάπτυξης συμμετέχει ή στην ομάδα που συνεργάζεται. Θα υπάρξει στις αρχές Μαΐου μία συνεδρίαση όπου θα συμμετέχετε με τους εμπειρογνώμονες και απλώς ήθελα να τονίσω αυτό το θέμα, ότι δηλαδή υπάρχει συμμετοχή. Ευχαριστώ. Η κυρία Λέβιν είναι καθοδόν. Οπότε ίσως θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, αλλά βλέπω ότι ούτε η κυρία Ζήμερη είναι εδώ. Τότε να προχωρήσουμε στο τελευταίο θέμα. Όχι, ήρθε εντωμεταξύ η κυρία Λόεβιν. Οπότε τώρα περνάμε στην παρουσίαση της κυρίας Λέβιν για, την, για το σχέδιο γνωμοδότησης για την κοινή ελευτική πολιτική κατόπιν προτάσεως της Ευρωπαϊκής ε, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για ε, την ε, ενιαία πράξη για την αλληλεία. Πρόκειται για μία απόφαση σε πρώτη ανάγνωση. Επιτρέπω στην κυρία Λέβη να καθίσει και να προετοιμαστεί. Της δώσουμε το χρόνο. Μην, μην βιάζεστε, δεν, δεν έχουμε πρόβλημα. Εσείς έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που μπήκα έτσι, αλλά ήμουν στην Επιτροπή Ιαλίας όπου συζητούσαμε το ίδιο θέμα. Οπότε... Μιλάμε για την αναδιάρθρωση και τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και αυτό γίνεται κατόπιν της προτάσεως για ένα νέο βασικό κανονισμό και φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι ήδη γνωρίζουν ότι η κοινή ε, αλληλευτική πολιτική δεν παρουσιάζει μία πολύ ενθαρρυντική εικόνα, μάλιστα θα έλεγα ότι είναι τραγική, γιατί έχουν μειωθεί σημαντικά τα αποθέματα αλίας στην Ευρώπη, ε, χάνουν το εισόδημά τους και οι Ευρωπαίοι αλληλείς, αλλά και περαιτέρω και πρέπει να βιαστούμε να επέμβουμε. Υπάρχει μία κοινή διαχείριση της Επιτροπής Αλληλείας η οποία έχει διάφορες πτυχές. Έχουμε από τη μία πλευρά της διμερής συμφωνίας για συμφωνίες συνεργασίας στον αλλιευτικό τομέα με διάφορες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, σε περιφερειακές οργανώσεις που διαχειρίζονται τον αλλιευτικό χώρο ε, για ε, μεταφερόμενα αποθέματα ε, αλληλείας τα οποία διαχειριζόμαστε και εμείς όπως ο τόνος και υπάρχει και η συνεργασία η οποία αναφέρεται εις την θαλάσσια διακυβέρνηση και τέλος υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δραστηριοποιείται με ιδιωτικές ε, επεμβάσεις στις υποανάπτυξη χώρες Και ένα άλλο θέμα για την εξωτερική διάσταση είναι ότι εισάγουμε ένα μεγάλο μέρος των ψαριών που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν του 60% των ε, ψαριών ε, εισάγονται όχι ε, όλα από τις ίδιες χώρες δηλαδή ο μεγαλύτερος εξαγωγός Προ προς την Ευρώπη είναι η Νορβηγία αλλά πολλά ψάρια έρχονται και από την Κίνα ε, και ε, ούτω καθεξής. Οπότε ε, βλέπουμε ότι ο απολογισμός είναι αρκετά θετικός και ένα βασικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τα αποθέματα τα αλληλευτικά ε, άνω του ελάχιστου βιώσιμου ε, προϊόντος δηλαδή ή ε, την απόδοση που μπορούμε να έχουμε αιώνια σαν να λέγαμε ένα επιτόκιο από τα ψάρια δηλαδή δεν πρέπει να μειώνεται το αρχικό ψυχικό σας κεφάλαιο διότι τότε όταν μειώνεται το κεφάλαιο θα μειωθούν όλα. Πρέπει να διατηρήσουμε το ανώτερο βιώσιμο απόθεμα και Γι' αυτό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Διότι όπως σας είπα, ε, μία από τις πιο βασικές αρχές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν μόνο αλευτικές συμφωνίες με χώρες οι οποίες ε, έχουν ε, επαληθευμένο πλεόνασμα ψαριών που μπορούν να μας πουλήσουν. Χρειάζεται Χρειάζεται λοιπόν καλή επιστημονική γνώση, να ξέρουμε ότι τα αποθέματα αυτά δεν έχουν τύχη υπερβολικής εκμετάλλευσης και αυτό έχει σχέση και με τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού. Όχι απλώς επιστημονικό πλεόνασμα που να λέει ότι δεν μπορούμε να ότι θα έχουμε ε, αλλιευτικά προϊόντα που δεν μπορούμε να αρέσουμε αλλά ότι θα μας προσφέρουν και τις αναγκαίες πρωτεΐνες και αυτό θα συνυπολογιστεί στο κόστος ε, του πλεονάσματος. Επίσης ε, εμείς είμαστε σύμφωνοι με την οικονομική αποζημίωση για την πρόσβαση στην αλληλεία που θα πρέπει να αποδεσμευτεί από τις ε, ενισχύσεις κάποιου τομέα δηλαδή όλα τα χρήματα χρήματα που πληρώνονται προς κάποια χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε δεν θα πρέπει να διατεθεί μόνο για την αλληλεία αλλά και για άλλες δραστηριότητες και να αποδεσμευτεί από αυτές ε, τις ε, ε, ενισχύσεις που δίδονται με σκοπό την ανάπτυξη κατά τρόπον ώστε να μην μειωθεί και το τμήμα της συμμετοχής ε, ε, παραδείγματος χάρη εάν πάρουμε την Γουινέα Μπισάου που έχει σημαντική αλλιευτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν μειωθούν τα αλλιευτικά της αποθέματα θα υπάρξει σημαντική επίπτωση στον προϋπολογισμό ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και αυτή είναι η ιδέα για την αποδέσμευση πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι Υπάρχει μία αποδέσμευση από την κατάσταση των αποθεμάτων. Η πρόταση δεν είναι πολύ αποτελεσματική όταν μιλάμε για υποχρεωτικές μεταφορές των λιευτικών αδειών και αυτό γίνεται για εσωτερική χρήση, για τα κράτη-μέλη και ε, όντως θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει ε, μία εμπορία αυτών των αδειών να προσπαθούν να αγοράσουν η μία την άλλη, να μην υπάρχει υπερβολική και πλεονάζουσα τονοχωρητικότητα, αλλά ε, θα πρέπει να, αυτό να μπορεί να ελεγχθεί και για άλλους τόλους πρέραν αυτό που ε, δραστηριοποιούνται στις διμερείς συμφωνίες κατά τρόπον ώστε οι μεταφερόμενες αλλιευτικές να μην μεταφέρεται σε πλοία τα οποία είναι ευρωπαϊκά και δραστηριοποιούνται εκτός Ευρώπη. Ε, αν υπάρχουν δηλαδή ιδιωτικέ συμφωνίες ή άλλου είδους συμφωνίες θα πρέπει αυτό να εξεταστεί και είναι πολύ βασικό γιατί στην πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέρευσε είδαμε ότι υπήρχε και μία ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία αφαιρέθη στη συνέχεια. Αλλά τώρα ξέρουμε ότι και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο στηρίζουν αυτή τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έτσι εγώ θα την επαναφέρω και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα με στηρίξουν. Υπάρχει και μία ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αλληλευτικές συμφωνίες οι οποίες επιδρά θετικά και η επέκτασή της θα πρέπει να ισχύσει και για τις αναθεωρήσεις της συμφωνίας του Κοτονού. Ε, αναφέρομαι εις ε, την ε, ρήτρα αποκλειστικότητος διότι είναι πολύ σημαντικό η υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να εξασφαλίσουν ότι εφόσον αλλιεύουν στην περιοχή εκείνη αυτό γίνεται βάσει των εγκεκριμένων αδειών και όχι εκτός κοινοτικού επίπεδου. Επιπλέον, προτείνω ορισμένες τροπολογίες σχετικά με τη διαφάνεια και η διαφάνεια βλέποντας τις τροπολογίες μία προς μία είναι ένας από τους στόχους που έχω θέσει για την κοινή αλλιευτική πολιτική να υπάρχει μία διάφανη πρόσβαση στην πληροφόρηση και αυτός είναι ένας από τους στόχους μας που είναι πολύ σημαντικός διότι ιδιαιτέρως ε, όταν πρέπει να καταρτιστεί ένα πλεόνασμα ε, των ε, υποθεμάτων αλίες πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτό προωθείται ε, και αντικατοπτρίζεται στις περιοχές όπου έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία αλληλευτική συμφωνία ε, διότι βλέπουμε ότι επιπλέον ενδέχεται οι χώρες αυτές να έχουν και ε, συμφωνίες με άλλες αλληλευτικές χώρες, στις Ηνωμένε Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα και αν δεν ξέρουμε πόσο ψάρι αλλιεύεται δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχει πλεόνασμα ή όχι και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρχει βάσιμα μία συμφωνία αλλιευτική. Ε, πρέπει επίσης να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει πόσο πληρώνει για κάθε αλλιευτική συμφωνία αλλά σε πολλές τρίτες χώρες όπου Υπάρχουν ε, διάφοροι ελευτικοί στόλοι, ούτε το Κοινοβούλιο δεν ξέρει ε, πόσες αλληλευτικές συμφωνίες υπάρχουν και τι πληρώνει κάθε χώρα για πρόσβαση ε, στην περιοχή. Έχω επίσης μία τροπολογία που αναφέρεται στην μεταφορά των αλλιευτικών αδειών διευκρινίζοντας ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να ισχύσει εκτός των υδάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, αρχικά ε, η Επιτροπή είχε πει ότι δεν πρέπει να ισχύσει εκτός των ε, κοινοτικών υδάτων και αυτό αναφέρεται και στην τροπολογία 3. για την τροπολογία 4. Λέμε ότι η εξωτερική διάσταση θα πρέπει να συνάδει με τις πολιτικές της ενώσεως στο τομέα του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης και του εμπορίου και να επιδιώκει τους ίδιους στόχους και να προωθήσει τα ίδια πρότυπα διαχείρισης της αλληλείας που ε, ε, εφαρμόζονται στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή οι επιχειρηματίες θα πρέπει να τα σέβονται, να σέβονται τις αρχές αυτές ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πρέπει να συνδυάσουμε ε, την εξωτερική αναπτυξιακή πολιτική με την εξωτερική αλληλευτική πολιτική για να υπάρχει μια καλή διακυβέρνηση. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό διότι διαπίστωσα ότι δεν είναι καθόλου επικοδομητική η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λέγει σε όλο τον κόσμο πόσο σημαντική είναι η βιώσιμη αλληλεία και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι άλλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία για να επιτύχουμε τους επιδιωκόμενους στόχους και των δύο πολιτικών και για να υπάρχει αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά την τροπολογία 5 που αναφέρεται στις ευθύνες των κρατών μελών δεν μιλάμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση των δικών τους επιχειρήσεων διότι το κράτος μέλος είναι αυτό το οποίο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες και αν τα κράτη-μέλη δεν συμμορφωθούν σε αυτές ε, τις διατάξεις θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ε, κυρώσεις ε, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο για χώρους εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πρέπει να υπάρχει κάπως μία δυνατότητα κυρώσεων. Και τέλος ε, υπάρχει ένας κατάλογος για να δούμε τι θέλουμε να διατηρήσουμε με τις βιώσιμες αλληλευτικές συμφωνίες, την έρευνα, την επιτήρηση, τη διαφάνεια και μία συνεκτική πολιτική στις τρίτες χώρες. Και τέλος, προς το τέλος υπάρχουν μόνο λίγες διευκρινήσεις ότι όλα αυτά πρέπει να αναφέρονται σε όλους τους στόλους. Στην τροπολογία 8 αναφερόμαστε στο θέμα της ε, σημαίας και της αλλαγής σημαίας διότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες εποφελούνται αλλιευτικών συμφωνιών επί έξι μήνες και μετά όταν εξαντληθούν οι ευκαιρίες με την αλλιευτική συμφωνία πηγαίνουν εις ε, μια άλλη χώρα και μετά συνεχίζουν να ψαρεύουν με την άλλη σημαία μέχρι να φτάσει 1η Ιανουαρίου που επανέρχονται στην κοινοτική σημαία πράγμα το οποίο είναι αντίθετο εις ε, την εκμετάλλευση του πλεονάσματος ψαριών και δεν θα έπρεπε να το ανεχθούμε. Τροπολογία 9. Την ανέφερα προηγουμένως. 10. Επίσης πολύ σημαντική διότι οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται για τις επιπτώσεις κάθε πρωτοκόλου προτού αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο πρωτόκαλο γιατί τώρα πολλές φορές αξιολογήσεις τις έχουμε εκ των υστέρων και όταν η αλληλεία έχει ξεκινήσει. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να έχουμε μια καλύτερη δυνατότητα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. σαν συνυπεύθυνοι μαζί με το Συμβούλιο για αυτές τις ε, συμφωνίες σχετικά με την τροπολογία 11. Μιλάμε για τους, τις επιχειρήσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος των ε, ε, ε, της προσβάσεως στην αλληλεία τώρα υπάρχουν σημαντικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις ενώ οι επιχειρήσεις πρέπει να καλύψουν το κόστος της πρόσβασης και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καλύπτει το κόστος για ορισμένες περιοχές. Ε, στην 12 φέρουμε πάλι στη διαφάνεια και στην τροπολογία 13 Νομίζω ότι με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων παρακολούθησης που παραχωρούνται στις μικτές επιτροπές δυνάμει των συμφωνιών βιώσιμης αλίας με τρίτε χώρε, η βοήθεια αυτή υπόκειται σε ανοιχτού χαρακτήρα και βάση λογοδοσία μηχανισμού επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένου διαθεσίμων μόνο στο κοινό λογιστικών ε, ελέγχων και ανεξαρτήτων αξιολογήσεων. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μία στήριξη του τομέα η οποία να είναι όντως ουσιαστική και δεν θα πρέπει η χρηματοδότηση να εξαφανίζεται χωρίς να υπάρχει μία τακτική αξιολόγηση. Λοιπόν, αυτά, αυτές ήταν οι τροπολογίες που είχα να κάνω και νομίζω ότι μπορώ τώρα να σας ευχαριστήσω και είμαι στη διάθεσή σας για τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μέσνερ. δεν περίμενα ότι θα μιλήσω τόσο σύντομα, αλλά σας ευχαριστώ που παρουσιάσετε λεπτομερώς το θέμα. Συμφωνώ με τις βασικές ιδέες γιατί βλέπω ότι ξέρει καλά την αλληλεία και όντως συμφωνώ γιατί οι προτάσεις αυτές είναι άξιες να στηριχθούν γιατί θα είναι σημαντικές για την αναπτυξιακή πολιτική ε, γιατί ε, η αλληλευτική η πολιτική δεν συμβάλλει μόνο στην διατροφική ασφάλεια αλλά και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας. Σκέφτομαι τη Σομαλία και άλλες χώρες οι οποίες έχουν τη βάση τους στην ανυπαρξία δυνατοτήτων. Δηλαδή η αλληλεία είναι ένα δυνητικό σημαντικό εισόδημα και γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Έχω παρατηρήσει ε, στις τροπολογίες οι οποίες πιστεύω ότι γενικώ για τους φιλελεύθερους είναι αποδεκτές και στην τροπολογία 3 αντιλαμβάνομαι ε, γιατί διατυπώσαμε διαβάσατε έτσι την τροπολογία αλλά βλέπω εδώ ότι στο άρθρο 28 μιλάμε για τις μεταφερόμενες ε, αρμοδιότητες αλλιευτικών αδειών και δεν ξέρω αν είναι κάτι όντως μεταφερόμενο και αν έτσι επιτυχάνουμε αυτό το οποίο επιζητούσαμε ή αν συνάδει με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά την τροπολογία 5 δεν βλέπω γιατί τα κράτη-μέλη ε, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση των επιχειρήσεων τους και πρέπει να αναλάβει τα διορθωτικά μέτρα η Επιτροπή. Ε, διότι εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορεί η Επιτροπή να εφαρμόσει αυτά τα οποία χρειάζονται και που πρέπει να προωθηθούν. Τώρα όσον αφορά τροπολογία 8, ε, νομίζω ότι η, η πρόθεση είναι να περιορίσουμε την αλλαγή σημαίας αλλά πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει για τα νέα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά ε, και ε, αυτοί οι οποίοι δεν λειτουργήσαν επί 24 μήνες με ευρωπαϊκή τη σημαία πρέπει να αποκλειστούν ή ποια λύση θα βρούμε. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες τροπολογίες νομίζω ότι είναι καλές και μπορούμε να τις δεχτούμε από πλευρά ε της, ε, των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. κύριε Κορτές ε, Λάστρα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με τις περισσότερες τροπολογίες και πάνω απ' όλα Συμφωνούμε εν γέννη με την πρόταση της Κομισιόν και σε ό,τι αφορά το μοντέλο ε, συμφωνίας για βιώσιμη αλληλεία στο μέλλον, την αλλαγή της ονομασίας, δηλαδή τρεις ε, είναι οι σημαντικές πτυχές. Πρώτα, είναι εξωτερική διάσταση και πρέπει να αποφεληθούμε ε, της στιγμής γιατί έχουμε την κοινή ελευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που όπως λέει και η εισηγήτρια είναι και προβεβλημένη και θετική και σε ό,τι αφορά τα λιεύματα και σε ό,τι αφορά τη βοήθεια προς τους πολίτες. Συμφωνούμε επίσης με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα διεθνή εργασιακά δικαιώματα. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, αλλά εν γέννη συμφωνούμε με τη μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών της ηγητρίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόγκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Και δεύτερον, θέλω να υπογραμμίσω δύο στοιχεία που πιστεύω ότι χρήζουν είτε τροποποίηση είτε διευκρίνηση στην πρόταση κανονισμού σε σχέση με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Πρώτο στοιχείο. Η απέτηση να ληφθούν υπόψη οι αναπτυξιακοί στόχοι κατά την εφαρμογή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και δεύτερον, είναι κάτι που υπογράμμισε σε τροπολογία της κυρία Λέβιν, για, τις για τη μεταβιβάσιμη αλία που δεν θα πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκά ύδατα. Έχω να καταθέσω τροπολογίες σε σχέση με αυτήν τη τροπολογία. Ο κύριος ε, Λάντμερ από την Κομισιόν τώρα έχει το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί ο συνάδελφό μου ουσιαστικά είναι αυτό ο οποίος ε, από τη διεύθυνση Β ε, εξωτερική ε, διάσταση από τη ΓΔ θα σας απαντήσει στα πιο πολλά ερωτήματα. Σύντομα, μια παρατήρηση την οποία είπα και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ. Ίσως υπάρχει μια μικρή παρανόηση για τις μεταβιβάσιμες συμβάσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα μέθοδο ώστε να μπορούν όχι οι Κομισιόν αλλά τα κράτη με έναν διαφορετικό νέο τρόπο να ρυθμίζουν και να παρακολουθούν την ίδια την πρόσβαση στην αλία. Εμείς λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουμε αυτή τη μέθοδο ίσως θα την έλεγα συνδιαχείριση ή αυτοδιαχείριση των αλληλευτικών ε, δυνατοτήτων, μια προσέγγιση δηλαδή η οποία θα επιτρέψει ευκολότερα και χωρίς χρήματα από τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο την καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ των διαθέσιμων πόρων και των αλληλευτικών δυνατοτήτων. Γιατί λοιπόν ε, αποκλείουμε τις συμφωνίες. Ε, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο οι συμφωνίες αυτές Υπάρχουν αλληλευτικέ δυνατότητε οι οποίε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση και μετά συμφωνία μεταξύ τη Ένωση και του τρίτου κράτου. Υπάρχει λοιπόν λόγο εξαίρεσή του. Εξαίρεση μάλλον των κρατών μελών την υποχρέωση να διαχειρίζονται τι αλληλευτικέ δυνατότητε κατά αυτόν τον τρόπο. Για τα γενικότερα για τα κοινοτικά ύδατα θεωρούμε ότι δεν είναι καλή ιδέα. Ε, ας δούμε τη Μεσόγειο. Όχι μόνο υπάρχει υπεραλίευση, αλλά εκεί που δεν υπάρχει δηλωμένη αποκλειστική ζώνη από τα κράτη-μέλη, ε, πλέον έχουμε να κάνουμε με διεθνή ύδατα μετά τα 12, για να μην πω και τα 6 μίλια. Άρα ε, τίθεται διαφορετικά το όλο θέμα. Και αυτό ε, είναι το πρώτο μου επιχείρημα. Το δεύτερο επιχείρημα, και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, είναι ότι ακόμη και στο Βόρειο Ατλαντικό, υπάρχουν πολλά αλλιευτικά σκάφη τα οποία δραστηριοποιούνται είτε σε ζώνες όπως ΝΑΦΚ, παραδείγματο χάρη, δηλαδή περιφερικών οργανισμών αλλιές και κοινοτικά. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε τη διάκριση. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο. Αν μου επιτρέπετε, λέει πρόεδρος, να δώσω το λόγο στον κύριο Αρσένη, που λίγο αργά βέβαια μου τον ζήτησε, και μετά θα σας δώσουμε το λόγο. Ε, να πω μόνο όπως είπε ο συντονιστής μας, ότι η κυρία Λόβινγκ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια αλλά θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε με πιο ενεργό τρόπο την παράνομη αλίευση και την υπεραλίευση. Έχουμε όλες αυτές τις συμφωνίες τις εταιρικέ για την αλληλεία και ταυτόχρονα έχουμε διάφορες ε, προβλέψεις για ποσά για την πρόσβαση στην αλληλεία. Ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο. Και ιδιαίτερα για τις χώρες γειτονίας. Κάποιες συμφωνίες οι οποίες θα μας επιτρέπουν να δίνουμε βοήθεια για να γίνονται σεβαστοί κοινοί κανόνες, οι δικοί μας κανόνες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Δεν είναι εύκολο στη Μεσόγειο να υπάρχει πρόσβαση στην αλληλεία πάντα. Και γι' αυτό στα πλαίσια της δεύτερης γενιάς αυτών των αλλιευτικών συμφωνιών θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης των ρυθμίσεων και κυρίως επιβολής των ρυθμίσεων, ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες όπως γύρω από τη Μεσόγειο και στα υπόλοιπα σύνορα της Ένωσης. Είναι μια ιδέα την οποία έχουμε συζητήσει αρκετά. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε και στη δική μας έκθεση. Δίνω το λόγο ξανά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ, θα αναφερθώ πάντα στις εταιρικές σχέσεις ε, συμφωνίες για την Αλία. Να ευχαριστήσω την κυρία Λέβιν καταρχάς. Διαπιστώνουμε μια ιδιαίτερη θα έλεγα σύγκληση με την εισηγήτρια για το σύνολο των προτάσεων της Επιτροπής. Αυτό αφορά και τα πλεονάσματα και τη μέγιστη αηφόρο ανάπτυξη και την αποσύζευξη, θα έλεγα, των δικαιωμάτων πρόσβασης και τις τομιακές διευκολύνσεις. Αυτό ισχύει επίσης και για τα θέματα της διαφάνειας και σε σχέση με τη σύνολη αλλιευτική δραστηριότητα, αλλά και σε σχέση με τις αξιολογήσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και διαφανείς. Ένα από τα θέματα που έχουμε μπροστά μας είναι το πώς θα εκφραστούν οι ιδέες αυτές και με ποιο τρόπο. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μία έχει παρουσιάσει μία ανακοίνωση και από την άλλη ένα βασικό κανονισμό, ο οποίος έχει γίνει δεκτός από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, θεωρώντας ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία πολιτικής φύσης και ορισμένα τα οποία είναι διακανονιστικής φύσης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν το πώς τώρα θα μοιράσουμε σωστά τους τομείς αυτούς έτσι ώστε να εντάξουμε όλους τους στόχους στο σωστό έγγραφο. Παίρνω το παράδειγμα για τον συντονισμό ανάμεσα στις αλλιευτικές συμφωνίες και την αναπτυξιακή πολιτική. Για μας αυτός είναι ένα σωστό στόχος που αφορά το σύνολο της πολιτικής της Ένωσης. Έχουμε και μια συμφωνία στη συνθήκη που αναφέρεται στα θέματα αυτά θα πρέπει να γίνει ειδικό στοιχείο αυτού του βασικού κανονισμού. Τίθεται σαν ερώτημα. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θέλουμε πλέον να εντάσσονται στο σύνολο των αλλιευτικών συμφωνιών. Το έχουμε επανειλημμένα πει. Έχει συμπεριληφθεί, όπως και άλλα στοιχεία, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του προηγούμενου Μαρτίου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα ειδικό άρθρο για μια αναγκαστική εφαρμοστική ισχύ στον βασικό κανονισμό. Γιατί βέβαια εμείς είμαστε στα θέματα της αλληλείας εντασσόμεθα και όχι στα θέματα της ανάπτυξης ούτε στα θέματα των διεθνών σχέσεων. Τίθενται λοιπόν τα θέματα αυτά. Θα ήθελα τώρα να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις λίγο πιο συγκεκριμένες για κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Πρώτον, θεωρώ ότι η πιο προβληματική για μας τροπολογία είναι η 11. Η 11 αφορά τον μακροπρόθεσμο λεγόμενο στόχο, ε, στα πλαίσια του οποίου το κόστος πρόσβασης σε αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να ε, πληρώνεται από ε, τις ωφελούμενες χώρες. Σε αυτή την περίπτωση τι θα μείνει από την αλλιευτική συμφωνία αν ο αλλιευτικός τόλος πληρώνει το σύνολο του κόστους της πρόσβασης. Θα υπάρχει το θέμα της διοίκησης, και της ανάπτυξης. Έχουμε ξεφύγει λίγο από τη λογική της εξωτερικής πολιτικής στον τομέα της αλίας. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει πράγματι τη φύση των συμφωνιών αυτών, την εμβέλεια των συμφωνιών αυτών και τον ελκυστικό τους χαρακτήρα. Γιατί ξέρετε ότι τα έσοδα τα οποία δίδουμε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στις χώρες αυτές είναι κάτι το εγγυημένο τώρα θα πληρώσουν οι εφοπλιστές. Αυτό εξαρτάται από μια ολόκληρη σειρά παραγόντων, από τη στρατηγική της αλίας. Δεν υπάρχει καμία σταθερότητα όμως, καμία ασφάλεια για την πληρωμή των ποσών αυτών, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεμπλακεί. Συνεπώς νομίζω ότι η δική μας συνεισφορά δίνει ένα κίνητρο στις τρίτες χώρες να υπογράψουν τη συμφωνία αυτή και να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης και διαχείρισης αλίας. Δεν έχουμε αυτό το ελκυστικό καρότο θα έλεγα για τη συνεργασία μας στην οικονομική και έτσι δεν θα τις βοηθήσουμε να διαπραγματευτούν μαζί μας κάποιες αλλιευτικές συμφωνίες οι οποίες είναι ένας τρόπος διαβελτίωσης της διαχείρισης των πόρων γενικότερα στα διεθνή ύδατα. Να προσθέσω ένα τελευταίο στοιχείο εδώ. Ο εξωτερικός στόλος είναι πολλαπλού χαρακτήρα. Έχουμε ένα στόλο ο οποίος αποτελείται από μεγάλα σκάφη με ισχυρά συμφέροντα. Έχουμε όμως και βιοτεχνική αλληλεία κοντά στις ακτές, το Μαρόκο, με πολύ μικρά σκάφη που δραστηριοποιούνται σε τομείς αλλιευτικούς, τους οποίους η αποδοτικότητα δεν είναι και πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με άλλους τομείς αλίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας προβληματίζει στην πρόταση αυτή και εδώ θα ήθελα να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να δείξει λίγο περισσότερη ευελιξία είναι το θέμα της αποκλειστικής ρήτρα. Αναφέρεται στο θέμα αυτό η τοπολογία 8, δεύτερο τμήμα. Η ρήτρα αυτή έχει σαν στόχο να επιτραπεί έτσι ώστε όλα τα ευρωπαϊκά σκάφη να αντιμετωπίζονται με τον κοινό τρόπο και κάτω από κοινέ συνθήκες εφόσον υπάρχει αλληλευτική συμφωνία η οποία είναι ενισχύ. Βλέπουμε βέβαια με ορισμένες χώρε, σαν παράδειγμα με την Καμπόν, ότι μπορεί να μην υπάρχει ε, τέτοιο ενεργό πρωτόκολλο. Όταν έχουμε τη ρήτρα αυτή αντιμετωπίζουμε ε, ένα διέξοδο. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν τα σκάφη και δεν μπορούμε να καταγγείλουμε τη συμφωνία αυτή με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο και μπλέκουμε σε μια κατάσταση έλλειψης δικαίου που δημιουργεί σε όλους πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι μια κάποια ευελιξία στα πλαίσια της εφαρμογής της ρήτας αυτής αποκλειστικότητας είναι σωστό να αναθεωρηθεί. Εδώ θα συμφωνήσω στο επόμενο θέμα με την κυρία Λέβενγκ. Εμείς έχουμε διευκρινίσει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να αποκλείσουμε αυτόν τον τουρισμό των σκαφών που αλλάζουν σημαία ανάλογα με τις συμφωνίες και ανάλογα με τις ποσοστώσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή όχι. Έγινε μία παρατήρηση σε σχέση με μία διατύπωση σημαντική. Αυτή λέγει ότι αν απαγορεύσουμε σε όλα τα σκάφη, όπως λέει η τροπολογία, τα οποία δεν είχαν σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν στην συμφωνία, ίσως να είναι ένα φράγμα στην είσοδο στη δραστηριότητα. Και αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι τα αλερετούρ, δηλαδή ε, μια σημαία κοινοτική που πηγαίνει στη σημαία του Μπελίζ και μετά ξαναγυρίζει όταν οι συμφωνίες είναι ευνοϊκές. Αυτές τις μετακινήσεις λοιπόν θα πρέπει να τις αποκλείσουμε, να τις αποφύγουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τις μορφές συνεργασίας που χρησιμοποιούσαμε και σε σχέση με το 24μηνο. Ένα τελευταίο στοιχείο για τις αξιολογήσεις. Όπως σας είπα είμαστε διατεθειμένοι να λειτουργήσουμε διαφανώς σε σχέση με τις αξιολογήσεις που είναι απαραίτητες πριν από την εκκίνηση κάθε διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι απαραίτητο. Είμαστε όμως και υπόλογοι σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα χρήματα στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών ιδιαίτερα για τα τομεακά κεκτημένα. Αλλά θα ήθελα κατά κάποιο τρόπο να κάνω μια προειδοποίηση σε σχέση με ένα πληθωρισμό ελέγχων, λογιστικών, αξιολογήσεων κτλ. Αν το κάνουμε αυτό σε όλες τις συμφωνίες όπως το προβλέπετε εσείς σε αιτήσια βάση, πιστέψτε με τότε δεν θα έχουμε χρόνο να κάνουμε τίποτα άλλο από το να διατυπώνουμε αξιολογήσεις και εκθέσεις. Ας προσπαθήσουμε να το δούμε το θέμα πιο σφαιρικά. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε αξιολογήσεις εξάντε και εξπόστο όταν συζητάμε μια τέτοια διαπραγμάτευση και να αποφύγουμε τις πληθωριστικές αυτές ελεγκτικές τάσεις. Και τελειώνω εδώ λέγοντας ότι σχετικά με τους εξωτερικούς λογιστικούς ελέγχους έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες. Δεν μπορούμε να στείλουμε εμείς το ελεγκτικό συνέδριο να πάει να ελέγξει τους λογαριασμούς ενός τρίτου κράτους, ανεξάρτητου κυρίαρχου συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο δαπάνησης των χρημάτων, σε σχέση με τους προσυμφωνημένους στόχους, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε λογιστικούς ελέγχους εμείς σε διοικήσεις χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε κυρία Λέβιν να αναδευτερολογήσετε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για την υποστήριξη. Το εκτιμώ όλους ιδιαιτέρως. Θα ήθελα να απαντήσω κάποια από τα ερωτήματα. Στην κυρία Μάισνερ να πω ότι ναι, έχετε δίκιο για τον τίτλο, θα πρέπει να το δούμε. Θα επανέλθω για την εξουσιοδότηση, η γιατί το ανέφερε και η Κομισιόν. Να ευχαριστώ τον κύριο Κορτές για την υποστήριξή του. Και περιμένω επίσης και τις τροπολογίες του κυρίου Πόγκα. Για τον Κρήτονα, σε σχέση με την παράνομη αλία, την άναρχη αδήλωτη αλία, το IUU λοιπόν αντιμετωπίζεται κυρίως ε, από τον κανονισμό περί ελέγχου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι εδώ το κατάλληλο μέρος. Ό,τι αφορά τώρα εταιρική σχέση χωρίς πρόσβαση σε αλίευση, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα. Η αποσύνδεση είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Διανοίγουμε δηλαδή ουσιαστικά εδώ νέους ορίζοντες. για το τι θα πρέπει να είναι ουσιαστικά εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα πρέπει να υπάρχει εξωτερική πολιτική χωρίς καν συμφωνίες ε, πρόσβασης. Δηλαδή μιλάμε για, όπως είπα, νέους ορίζοντες. Αλλά θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Επομένω, ε, για να έρθω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με έχει λίγο ε, μπερδέψει αυτό που είπε ο πρώτο ομιλητή για αυτέ τι μεταβιβάσιμε αλλιευτικέ παραχωρήσει ότι είναι κάτι εσωτερικό. Εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν θέλετε να επιβάλλετε εσείς κάτι. Δηλαδή, αν ένα σκάφος ε, έχει τη σημαία ενός κράτους μέλους και το κράτος μέλος πρέπει να υιοθετήσει αυτό το σύστημα για όλα τα σκάφη πάνω από 12 μέτρα, όλα τα σκάφη, ακόμη και αν δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να περιληφθούν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται ακριβώς. Ποια είναι η πρόθεση της Κομισιόν. Όλα τα σκάφη εκτός που δραστηριοποιούνται εκτός ε, των αλληλευτικών ε, συμφωνιών να πρέπει να περιληφθούν. Αν είναι ναι, εμείς είμαστε κατά. Δεν νομίζουμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει παγκόσμια αυτό το σύστημα μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων, γιατί αυτό θα είναι εντελώ αρνητικό για τι αναπτυσσόμενες χώρες, διότι οι μεταβιβάσιμες αλλιευτικές παραχωρήσεις βασίζονται σε ιστορικά αλλιεύματα και οι αναψώμενες χώρες βέβαια έχουν ήδη θεσπίσει τις αλλιευτικές του παραχωρήσεις παγκοσμίω ε, με βάση, αν θέλετε, την οικονομική ανωτερότητα, την οικονομική δύναμη. Το να έχουμε λοιπόν τώρα να θεσπίσουμε παγκόσμιο ε, σε ένα σύστημα μεταβάσεων αλληλευτικών παραχωρήσεων για τις αναπτυσσόμενες χώρες, νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές τις χώρες αν θέλουν να αγοράσουν εντό αγωγικών κάποια λεφτική παραχώρηση. Για τα άλλα σχόλια της Κομισιόν. Ε, με εκπλήσει κάπως με εκπλήσουν μάλλον τα σχόλια. Δηλαδή, αν η λευτική βιομηχανία πληρώσει το δικό τη μερίδιο, δεν καταλαβαίνω πώ με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουν ε, πραγματικά βιώσιμη αλληλεία, ένα πραγματικά βιώσιμο αλληλευτικό πλαίσιο για του Ευρωπαίου, αλληλεία που δραστηριοποιούνται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνω και δεν βλέπω το λόγο. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποσκοπεί στο να πλαισιώσει του ε, παράγοντε οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκτό υδάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να σέβονται και αυτοί και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα για τροφή, το πλεόνασμα των ε, ε, ψαριών να μην συνεισφέρουν δηλαδή στην υπεραλίευση κάποιων ειδών κτλ. Όλα αυτά με στόχο να έχουμε ένα πιο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Για πολλές χώρες γνωρίζουμε ότι ο ελευτικός τομέας, ο ελευτικός κλάδος μάλλον, εκφράζει παράπονα γιατί ε, σε αυτά τα ύδατα ε, δεν υπάρχουν... Ε, αυτές οι προτάσεις που θα επέτρεπαν να υπάρχει ένα ασφαλές ε, πλαίσιο λειτουργίας. Δηλαδή μείωση φορολογίας του καυσίμου, και κάποιες άλλες εξασφαλίσεις. Και σε ό,τι αφορά τα, το γνωμοδοτικό συμβούλιο μακράς στο το LDRAC, έχει κάνει ένα έχει κάνει μια δήλωση με την οποία συμφωνεί ότι οι θα πρέπει να πληρώνουν ένα θεμητό ε, μερίδιο του κόστους. Άρα δεν νομίζω ότι είναι κάτι επίμαχο. ούτε για τους ίδιους τους αλληλείς και δεν νομίζω ότι μειώνει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τη βιώσιμη αλληλευτική πολιτική σε άλλους χώρες. Σε ό,τι αφορά αυτή την τροπολογία για την αλλαγή σημαίας, ναι, βέβαια θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσαρμογές προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Αλλά για να απαντήσω τώρα στην κυρία Μάισνερ, δεν νομίζω κατά βάση ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε νέα σκάφη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της συμφωνίας. αν αυτό μπορεί να είναι εμπόδιο δηλαδή για την ε, εισαγωγή νέων σκαφών. Δεν θα μπορεί να το κάνει ο ε, αλλιέας ή τέλος πάντων η επιχείρηση. ναι να μεταφέρουν τις να δυνατότητες, αλλά όχι να εισαγάγουν νέα σκάφη, νέα πλοία. Θα το εξετάσω πάντως, δεν ξέρω αν ε, μήπως μπορούσα να το τροποποιήσω κάπως. Για τη ρήτρα ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτική συνοχή κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, πρόβλημα με το να μπει αυτή η ρήτρα στη, στο βασικό κανονισμό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάπου υπάρχει μια απόφαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική συνοχή, συνέπεια κτλ. Και, και από εκεί πέρα δεν πρέπει να αναφέρεται. Δεν θα πρέπει, νομίζω, να το να πάψουμε να επαναλαμβάνουμε αυτή την πολύ καλή αρχή. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδότης. 8 Μαΐου, 12 το μεσημέρι. Λίγη προθεσμία. Και τώρα περνάμε σε ανταλλαγή απόψεων για την γνωμοδότηση της συναδέλφου Γκάμπι Τσίμερ. Τροποποίηση του παραδείγματος 1 του κανονισμού 1528 του Συμβουλίου. Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Η εισηγήτρια είπα είναι συναδελφός μας η κυρία Τσίμερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με τον κανονισμό αυτό του 2007 1528 ε, κάθετος 2007 ε, έχουμε ένα κείμενο το οποίο δεν είναι μόνο προβληματικό αλλά νομίζω ότι εδώ και η Επιτροπή και η, το τμήμα εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν όσον αφορά την ε, πρόταση για την ε, τροποποίηση του παρατήματος γιώτα ε, του κανονισμού 1528-2007. Υπάρχουν μέλη που ήταν εδώ και στην προηγούμενη θητεία και ίσως θυμούνται πόσες συζητήσεις είχαν γίνει το 2007 όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μεγάλη μεγάλες πιέσεις, εξίσχυσε μεγάλες πιέσεις στις χώρες ΑΚΕΙ για να μπορέσει να καταλήξει κάπου στο τέλος του 2007. Είχαμε τότε συμφωνήσει ότι θα υπήρχαν προσωπι... προσωρινές συνθήκες για να μπορέσει να εξασφαλιστεί εντωμεταξύ η ε, ε, πρόσβαση στην αγορά αλλά είχαμε ήδη πει ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι συνθήκες αυτές είχαν βασιστεί εις ε, τα ουσιαστικά θέματα μόνον και θα έπρεπε να υπάρχουν και τελεσίδικες συμφωνίες και αυτό είναι κάτι σαφές διότι εάν ε, λάβουμε υπόψη μας ότι ε, οι διαπραγματεύσεις για μια συνθήκη είναι μια μακριά διαδικασία και για τους δύο εταίρους που οδηγούν σε θέματα υπαρξιακά και ε, τραβάν εις μήκος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Επιτροπή αναπτύξεως δεν πρέπει να δεχθεί οι χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ε, συνάψει μία συμφωνία ή την έχουν κυρώσει αλλά δεν θα την έχουν εφαρμόσει μέχρι το τέλος του 2013 ή την έχουν κυρώσει, δεν την έχουν κυρώσει αλλά ούτε καν θα την έχουν κυρώσει ως το τέλος του 2013 θα πρέπει να αποκλειστούν από την, ε, την πρόσβαση στην αγορά. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για την θέση της Επιτροπής Ανάπτυξης για να υπάρχει μία συνεκτική πολιτική η οποία θα μπορέσει όντως να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης αυτών των χωρών και να μην δημιουργήσει αντιφατικές προωθήσεις εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τελικά εδώ δεν πρόκειται μόνο για υπαρξιακά προγράμματα διότι οι χώρες ε, ε, ε, LDC έχουν προβλήματα και οι άλλες χώρες οι οποίες, μάλλον οι φτωχές χώρες θα είχαν σημαντικά προβλήματα οι μέσου εισοδήματος χώρες και αυτές θα είχαν προβλήματα και εμείς επιζητούμε κατά βάθο να υπάρξει ε, μία διαπραγμάτευση ε, για τα θέματα αυτά και ορισμένα ευαίσθητα ε, εξαγωγικά προϊόντα να δούμε ότι δεν καλύπτονται εδώ για το βόλιο ε, ε, και τα οποροκυπεστικά όπως και άλλα. Γι' αυτό το λόγο η πρόταση δικιά μου είναι στη γνωμοδότησή μας προς ε, την Επιτροπή Εμπορίου η οποία ηγείται και πρόκειται να καταρτήσει την εισήγηση να ζητήσουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψουμε αυτή την τροποποίηση του κανονισμού γιατί θεωρώ ότι δεν είναι σωστό τα υποανάπτυξη κράτη, ε, η διαπραγματευτική έτερη μας, ε, η οποία ε, θα χρειαστεί να βρεθούν υπό τέτοια πίεση και αυτό είχε ήδη επισημανθεί όταν έγινε η πρώτη διαπραγμάτευση το 2007 ότι δεν μπορεί κανείς να πιέσει σε τέτοιο βαθμό τα κράτη και να ε, να υποστούν μία πίεση την οποία δεν μπορούν να αντισταθούν. Επίσης είχαμε τονίσει τότε και αυτό σημαίνει ότι είναι βασικός λόγος ότι σαν Επιτροπή Ανάπτυξης δεν θα δεχθούμε μία τέτοια τροποποίηση του κανονισμού διότι για την περιφερειακή συνεργασία των χωρών και θα σημάνει μία μεγάλη περικοπή διότι αν το ένα κράτος έχει υπογράψει το άλλο όχι, τα τρίτα κράτη πρόκειται να σκεφτούν πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν επηρεάσει την ε, περιφερειακή αλληλεγγύη και την ε, ε, περιφερειακή διασύνδεση αυτών των χωρών και δεν είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε. Είχαμε μάλιστα προειδοποιήσει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές και πιστεύω ότι αυτό είναι το σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε και προτείνω στην Επιτροπή μας ε, να ζητήσουμε από την Επιτροπή που ηγείται να απορρίψει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Τσίμα για μια συνολική εξέταση της κατάστασης που δημιουργείται από την έκθεση αυτή. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ίσως εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινώντας θα ήθελα να μάθω αν μπορεί να επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι χώρες μέσου εισοδήματος θα ενταχθούν στα πλαίσια αυτού του GSP. Υπάρχουν ε, διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου, αλλά μου λέγουν ότι αυτή είναι η πιο πιθανή κατάληξη. Και αυτό μας οδηγεί σε μια κατάσταση ε, η οποία θα έλεγα χαρακτηρίζεται από σύγχυση. Εάν δεν γνωρίζουμε πλήρως τι θα γίνει στις μέσες λεγόμενες χώρες, μέσω εισοδήματο, στην ουσία παίρνουμε αποφάσεις για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε ε, τι θα δημιουργήσει. σχετικά με τους κανονισμούς για την πρόσβαση στην αγορά. Ανησυχώ για την κατάσταση στην Ποτσουάνα και στην Αμίμπια, για τη θέση στην οποία βρίσκονται οι δύο αυτές χώρες, οι οποίες θα ενταχθούν πιθανώς σε αυτές τις ε, μέσου εισοδήματος αλλαγές στην GSP. Νομίζω ότι οι χώρες αυτές οι δύο είναι ένα καλό παράδειγμα για το ε, τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε εμείς σαν ύπασμοι που δεν ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία όπως υποτίθεται, αλλά δημιουργεί προβλήματα επιπλέον. Η Μποτσουάνα και η Ναμίμπια ε, ε, είναι σε τελωνιακή ένωση με την Νότια Αφρική για πάρα πολλά χρόνια και ο λόγος για τον οποίο δεν θέλουν να προσυπογράψουν σε ένα ΙΠΑ είναι ότι η Νότια Αφρική δεν το κάνει. Και υπογράφοντας ένα τέτοιο πρόγραμμα με τις άλλες χώρες του νοτιού τμήματος στην Αφρική, τότε για, για πρώτη φορά δεν θα είναι σε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Νότια Αφρική, με την οποία έχουν πολύ στενές σχέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι διόλου ικανοποιητική. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε οι χώρες αυτές, γιατί η Νότιος Αφρική από ό,τι καταλαβαίνω έχει μια συμφωνία εμπορική με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σειρά της και αυτό πιθανό θα οδηγήσει ίσως και σε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Οπότε τι θα γίνει με την Αμίμπια και την Μποτσουάνα. Θα βρεθούν εκτός όλων των συμφωνιών και στην ουσία θα μείνουν μόνες τους και χωρίς κανένα ιδιαίτερο μέσο. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βέβαια κατανοώ τις ανησυχίες τους εφόσον δεν υπάρχει προθεσμία, τότε θα υπάρξει πιθανότητα σύγκρουσης με τους κανόνες του ΠΟΕ. Και κατανοώ επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αυτές οι οποίες πήραν τη δύσκολη απόφαση να υπογράψουν ένα ΙΠΑ, όπως χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, ότι το κάνουν κάνοντας και ορισμένες θυσίες και με ενοχλεί γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια αναβολή ε, για τη διαδικασία αυτή στην Αφρική. Δεν είμαι βέβαιος βέβαια ε, ε, για το ότι η σωστή απάντηση είναι η πλήρης απόρριψη. Αυτό όμως που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι διόλου ικανοποιητικό. Και διαρωτώ με αν μια συμβιβαστική λύση θα ήταν να πούμε ότι θέλουμε εμείς η προθεσμία αυτή για τη συμφωνία στην πρόταση πρόσβαση στις αγορές να παραταθεί μέχρι το 2016. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία ακούγεται, τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Βάλλη ίσως. ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους βουλευτές ε, που έδωσαν ε, τις απόψεις τους για αυτό το θέμα. Θα ήθελα, εν συντομία, να σας θυμίσω το πλαίσιο, αυτό το βιβλιαράκι που σας δείχνω, Συμφωνία Κοτονού δηλαδή, που υπογράψαμε το 2000, δηλαδή πριν από 12 χρόνια. Στη Συμφωνία του Κοτονού θεσπίζεται αυτό το κοινό πλαίσιο με τις χώρες ΑΚΕ για τη διαπραγμάτευση και την υλοποίηση Συμφωνιών Οικονομικής ε, εταιρική Σχέσης. Μετά, αφού διάβασα μάλλον την, ε, το σχέδιο έκθεσης, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι απλά στόχος η συμβατότητα ε, με τον ΠΟΕ. Μιλάμε πιο πολύ για εμπορικές εταιρικές σχέσεις με στόχο την ανάπτυξη. Γιατί το εμπορικό καθεστώς έδειξε ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των λαών των χωρών για του οποίου προοριζόταν. Θέλουμε λοιπόν να διαπραγματευτούμε αυτές τις συμφωνίες και ναι πράγματι ε, δεν μπορεί να πει ε, ότι θα δια... μάλλον μπορεί κανείς να πει θα διαπραγματευόμαστε εφαόριστον. Ε, δεν είναι και τελείω ε, παράλογο αυτό, ιδίω για την πρώτη πενταετία των διαπραγματεύσεων ή τα πρώτα δέκα χρόνια των διαπραγματεύσεων. Αλλά μετά από 10 χρόνια λοιπόν, αφού το ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα μια κατάσταση όπου είπαμε να μην το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, Είπαμε, θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2007. Στο πλαίσιο της περίοδου αυτής θα διαπραγματευτούμε αυτές τις συμφωνίες. Πετύχαμε κάποια αποτελέσματα, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για υλοποίηση την 1η Ιανουαρίου του 2008. Και ακριβώς αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλόπιστα ε, έχει προτείνει αυτή τη μεταβατική διευθέτηση που είναι ο κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά με στόχο να γεφυρώσει ε, το σύστημα των εμπορικών προτιμήσεων κοτονού και το νέο ε, συνολικό καθεστώς των συμφωνιών εταιρικής, οικονομικής εταιρικής σχέσης. 36 δικαιούχοι του κανονισμού, οι 18 έχουν περάσει τη γέφυρα, υπάρχουν άλλοι 18 όμως εταίροι που δεν σημείωσαν επαρκή πρόοδο ακόμη Παρ' όλα αυτά όμως υποφελώνται των ίδιων πλεονεκτημάτων με τους 18 που έχουν πλέον πλήρη πρόσβαση στην αγορά μας. Και αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε είναι δίκαιο από ε, νομικής πλευράς, αλλά ούτε και γενικότερα δίκαιο το θεωρούμε στο πλαίσιο των χωρών εκεί, αλλά και απέναντι και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες ζητούν ε, καλύτερη ή ελεύθερη πρόσβαση για τις αγορές μας και βλέπουν ότι κάποιοι φαίνεται να μην υποβάλλονται σε κανέναν περιορισμό. Το σχέδιο γνωμοδότησης αναφέρει τη σημασία των επενδύσεων για την ανάπτυξη. Ο αναπτυξιακός στόχος, εμπόριο, επενδύσεις, αυτά είναι μια καλή βάση και ο κανονισμός για την πρόβληση στην αγορά κατά την άποψή μα δεν μπορεί να επιτύχει αυτό το σκοπό. Πρέπει λοιπόν το συντομότερο να αντικατασταθεί με κάτι πιο στέρεο, που θα είναι και πιο δίκαιο και συνολικότερο από πλευράς αναπτυξιακή πολιτικής. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έξω και δεν προτείνουμε η τροποποίηση αυτή να εφαρμοστεί είτε τη μέρα της έγκριση τη είτε την επομένη, αλλά έχουμε θέσει ω προθεσμία ε, το 2014. Έξι χρόνια λοιπόν από θέση ίσχυ του κανονισμού. Ο αντίκτυπος νομίζουμε ότι μπορεί ε, να είναι εντελώ διαχειρίσιμος ε, εξαρτάται από την απόφαση των πλεκομένων χωρών και νομίζουμε ότι είναι λογικό να ζητήσουμε αυτή τη στιγμή τα κράτη να, είναι, να τηρήσουν μια αποφασιστική στάση σε σχέση με τις συμφωνίες που έχουν εγκρίνει και σε σχέση με τις επαγγελματίες που κυρίζονται το 2002. Merci beaucoup. Euh, la parole... Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε το λόγο? Ναι, θέλω το λόγο. Ε, δεν απάντησε την ερώτησή μου η Κομισιόν για την Ναμίμπια. Γρήγορα. Ναι, να σας ζητήσω συγγνώμη που το ξέχασα και μπορώ να σας πω ότι οι χώρες οι οποίες είναι στην κατηγορία αυτή του συγκεκριμένου εισοδήματο ε, για τρία χρόνια δεν θα ε, εποφελούνται πλέον ε, του GSP. Εσείς αναφέρατε την Ναμίμπια και άλλη μια χώρα. Δύο χώρες που ενδεχομένω να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Μεταξύ των 36 είναι οι δύο μόνες χώρες. Αυτό που δεν ε, μπορώ εύκολα να δεχθώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί πρόβλημα στην περιφερειακή ολοκλήρωση. Πρέπει να σα θυμίσω ότι η Νότια Αφρική έχει συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1999, ανεξαρτήτως του ότι Αυτό συζητήθηκε. Μία χώρα αποφάσισε να διαπραγματευτεί και να υπογράψει και οι δύο πάντως αποφάσισαν να διαπραγματευτούν τις συμφωνίες. Not sustainably... Αλλά ε, δεν μπορεί να υπάρξει μια βιώσιμη βάση για αυτές τις ε, συμφωνίες. Το θέμα είναι αυτές οι χώρες ε, τι θέλουν να κάνουν με αυτές τις συμφωνίες. Είναι θεμητό αυτό που θέλουν. Η Νότια Αφρική είναι σε μια πιο άνετη θέση γιατί οι προτιμήσεις τους δεν θα εξαρτηθούν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 Für mich gibt es darüber hinaus noch eine ganze andere Reihe von weiteren Fragen, die jetzt leider ebenfalls. Έχω και άλλα πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη και τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν. Δηλαδή γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει απαιτήσει οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ ε, τους κανόνες που συνάδουν με τους ε, ε, με την νομοθεσία του ΠΟΕ. Δηλαδή προβλέπεται ότι πρέπει να μειωθούν ε, τα, ε, οι δασμοί για μία σειρά προϊόντων. Πρέπει να υπάρχει μία ευελιξία από τα εμπλεκόμενα κράτη και αυτοί οι ίδιοι αμφισβητούν ότι δεν μπορούν πλέον να διαπραγματευτούν κάτι και γιατί μία χώρα σαν την αιτή η οποία έχει τόσο υποφέρει λόγω του σεισμού και της καταστροφής που προκάλεσε γιατί ακόμη και μία τέτοια χώρα θα πρέπει να εξαιρεθεί από το παράρτημα ένα. δεν είναι δυνατόν να πρέπει να μετρούμε ε, να μην μετρούμε, να μετρούμε όλους με τα ίδια μέτρα και σταθμά και αν θέλουμε να υπάρξει μία ανάπτυξη αν θέλουμε να συνεχίσουν να αναπτύσσονται οι χώρες και να έχουμε εταίρους στην αγορά και να υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είπαμε ότι ορισμένοι συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα αλλά δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να, να φερθούν σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία σαν καταληκτική και μετά να υπέρθει το χάος. Δεν μπορεί να πιέζει κανείς τα κράτη αυτά που αντιμετωπίζουν ήδη τόσες δυσκολίες και να τους λέμε ότι εσείς δεν, έχετε, δεν θεωρείστε ισότιμοι εταίροι για μας. Ε, το ίδιο θέμα υπάρχει με την ε, Ναμίμπια και την Μποτσουάνα. Τα ίδια θα μπορούσαν να λεχθούν και για άλλες χώρες της Αφρικής. Υπάρχουν παραδείγματα ή διάφορα πρότυπα. Ε, αν παραδείγματο χάρη δέχεται κανείς από όλη την Ανατολική Αφρική μόνο την Κένια. Ε, και, δεν, και απορρίπτει όλους τους εταίρους από την ε, περιοχή αυτή. Ε, τι θα γίνει, θα υπάρχουν καταστροφικές επιπτώσεις για τις εμπλεκόμενες χώρες και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συνυπολογιστεί στις διαπραγματεύσεις και τελικά δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Εγώ λοιπόν εμένω Θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση ε, του κανονισμού μου ε, από το 2014 ε, δεν θα επιτρέψει μία συνεκτική ανάπτυξη, δεν θα επιτρέψει μία δίκαιη συνεργασία η οποία θα εφαρμόζει τους κανόνες του ΠΟΕ και που θα καθιαστεί στη δυνατόν οι χώρες αυτές να προοδεύσουν. Θα πρέπει λοιπόν να προτείνουμε ε, στην ε, Επιτροπή Εμπορίου να μην δεχθεί την τροποποίηση αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τσίμερ. Σας υπενθυμίζω ότι η αποδοχή ή όχι αυτή της συμφωνίας θα αποφασιστεί με την ψηφοφορία 14 Μαΐου στην επόμενη συνεδρίαση και τελευταίο θέμα σήμερα είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή του Σαχέλ. Όπως ανεφέρθη στην αρχή έχουμε εδώ τον κύριο Σέσβι Τεγκρού ε, επικεφαλής εις ε, την Γενική Διεύθυνση για την περιοχή της Ανατολικής Αφρικής και του Ινδικού ωκεανού και έναν ακόμη προσκεκλημένο ο οποίος θα παρουσιάσει τα διάφορα θέματα και τις λύσεις που προτείνουν. Εγώ σαν μόνιμος εισηγητής αυτής της Επιτροπής για την ανθρωπιστική βοήθεια θα παρουσιάσω τα θέματα διότι πήγα πριν από ένα μήνα στο Τσάντ, στην περιοχή του Σαχέλ ε, και ευχαριστώ την ΕΚΟ και την Αντζεμίνα για την πολύ συμπαθητική οργάνωση της αποστολής, διότι οι χώρες του Σαχέλ πάσχουν από ε, μόνιμο υποσυτισμό εδώ και 10 χρόνια και τώρα η κρίση αυτή προσωμιάζει σε αυτήν του 2010 οι κακές εσοδίες του 2011, η αύξηση των τιμών των ε, τροφίμων, ε, ε, η καλπάζουσα δημογραφική αύξηση, η φτώχεια εξηγούν την κρίση και γι' αυτό πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα πέντε κράτη από τα πιο σοβαρά που πλήγησαν πιο σοβαρά έχουν ζητήσει την διεθνή συνεργασία και έκαναν έκκληση γι' αυτό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε την ε, ε, ανεπάρκεια τροφίμων και ορισμένες χώρες έχουν ξεκινήσει με δωρεές. Η κρίση ε, γίνεται πιο σοβαρή, δεν επαρκεί η διεθνής βοήθεια και πρέπει να δράσουμε πολύ γρήγορα. Θεωρούμε ότι 15,5 εκατομμύρια άτομα πλήττονται από αυτή τη διατροφική κρίση. Πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά θα πεθάνουν από σοβαρό υποσυτισμό εάν δεν ενταθούν άμεσα τα μέτρα. Διότι ο υποσυτισμός πλήττει τα παιδιά και επιπλέον δημιουργεί αμετάκλητες επιπλοκές και ο υπεύθυνο της UNICEF θα μας ενημερώσει. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την διατροφική ασφάλεια ε, στο πρόγραμμα ανάπτυξης ε, όσον αφορά την κατάσταση του Μαλή. Η ασφάλεια επιδεινώνεται, οι Τουαρέγ έχουν υποφεληθεί. Ε, από το στρατιωτικό πραξικόπημα και στο Ισλαμικό Μαγκρέπ αυξάνεται η επιρροή τους όπου υπάρχει και σοβαρό εμπόριο ναρκωτικών και το Μαλί συγχρόνως αντιμετωπίζει μία σοβαρή διατροφική κρίση και είναι μία από τις ε, πιο σοβαρά ε, πληττόμενες χώρες του Σαχέλ. Μπορεί δε η κατάσταση αυτή να επεκταθεί και στις γειτονικές χώρες γι' αυτό και δεν ε, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να βοηθήσουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν 136.000 πρόσφυγες στις ε, γειτονικές χώρες, τον Μπουρκίνα Φάσο, την ε, Αλγερία και τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να ενισχύσει την βοήθεια βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ε, ανάπτυξη του Σαχέλ. Όπως σας είπα ήμουνα σε αποστολή στο Τσάντ, στο Σανέμ. Δεν ξεχάσαμε την κρίση αυτή, αλλά η προσοχή ε, της ε, κοινή γνώμης δεν επαρκεί δεδομένων των αναγκών, δεν υπάρχει επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια στο Τσάντ ε, και υπάρχει 20% υποσυτιζομένων ατόμων ε, και έχουμε πολλούς πρόσφυγες οι οποίοι γύρισαν στο Τσάντ λόγω της κρίσης στο Μαλί διεκόπησαν οι είσοδοι εμβασμάτων ε, και αυτή τη στιγμή το Τσάντ έχει κάποια ασφάλεια και δεν εμποδίζει πολιτικά την ανθρωπιστική βοήθεια, πράγμα που δεν ισχύει για άλλες χώρες όπου ε, ε, ε, υπάρχει γενικό συναγερμός. Η ομάδα Μπόκο η στο Μαλί και άλλοι οργανισμοί επεμβαίνουν. Δεν υπάρχει κανένα επίγον πρόγραμμα δράσης, δεν υπάρχει δυνατότητα επενδύσεων και η χώρα έχει εισοδήματα από το πετρέλαιο και έχει ένα δηληστήριο το οποίο ε, συνδιαχειρίζεται με τους Κινέζους ε, διαπίστωσα όταν συνάντησα τον Υπουργό Γεωργίας ότι ε, ο ίδιος Υπουργός είχε έρθει ε, να παρουσιάσει τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς να έχει να προτείνει καμία στρατηγική λύση. Υπάρχει λοιπόν μία σοβαρή ανθρωπιστική κρίση πέραν αυτού και στο κέρας της Αφρικής και στο στη Βόρειο Κένια και ό,τι είδα στο Τσάντ πραγματικά με σόκαρε διότι το 2012 στην, σύμφωνα με την ε, UNICEF 126.000 μόρα θα πληγούν ε, από σοβαρό υποσυτισμό ε, επισκέφθηκα μία περιοχή και στις οάσεις είδαμε ότι πρέπει να υπάρξει προστασία και προσωπικά με εξέπληξε η έλλειψη ε, εμπειρου προσωπικού της ΦΑΟ. Για να μην υπάρξει λοιπόν μία νέα επισητιστική κρίση θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητα αντοχής των ε, πληθυσμών και ε, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη της περιοχής και για να μπορέσει να, να να είναι αποφασιστική η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συσφίξει τις σχέσεις με το Τσάντ που μπορεί να βοηθήσει τον πληθυσμό για να μην πεθάνει. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 8 με 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν χρειάζομαι 10 λεπτά γιατί αυτά τα οποία είπατε είναι σαφή και επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις που κάνουμε εμείς για την κατάσταση στο ΣΑΕΛ και ειδικά στο Τσάδ. Να σας ευχαριστήσω για την αποστολή σας. Είδαμε με χαρά ότι γνωρίζετε πλέον από κοντά τις δυσκολίες του πληθυσμού και των ανθρωπιστικών οργανώσεων να εργαστούν σε χώρες όπως το Τσάρ. Το Τσάρ δεν είναι τόσο ανασφαλές όσο ο Νίγηρας και το Μαλί. Οι συνθήκες εργασίας σε άλλες χώρες της περιοχής του Σαχέλ είναι χειρότερες από το Τσάρ. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε στο Σαχέλ σήμερα είναι η ε, μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που σοβεί σήμερα. 55 εκατομμύρια θίγονται άμεσα. Οι προσπάθειες της Επιτροπής και της ΕΚΟ προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες 8 εκατομμυρίων από τα 55 που είναι υψηλό ποσοστό αλλά αφήνει 7 εκατομμύρια, από τα 15 συγγνώμη, αφήνει 7 εκατομμύρια ακάλυπτα. Η συζήτηση σήμερα το απόγευμα νομίζω είναι πάρα πολύ εύθετη γιατί αντιμετωπίζουμε εκκλήσεις για περαιτέρω χρηματοδότηση από πλευράς των διεθνών οργανισμών και των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, ζητούν επιπλέον χρήματα, ζητούν να υπάρξει μια διάσκεψη για κινητοποίηση της ε, διεθνούς προσπάθειας. Εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό ήδη από το μήνα Φεβρουάριο, στα πλαίσια της ομάδας επαφής με, τις, ε, με τους ε, εταίρους, τους διμερείς εταίρους και τα Ηνωμένα Έθνη. Είπατε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, βλέπετε όμως ότι μέχρι τώρα η διεθνής απάντηση στην κρίση είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να κινητοποιήσουμε την βοήθεια που χρειάζεται. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακράν ο μεγαλύτερος δωρητής που καλύπτει ανάγκες στο Σαχέλ. Έχουμε τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή, αλλά ζητάμε τη διεθνή κοινότητα να μας ενισχύσει, γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας που είναι 750 εκατομμύρια που ζητούνται από το Ηνωμένα Έθνη, είμαστε στο 40% του ποσού αυτού. Εμείς πήραμε τα μαθήματά μας από το κέρας της Αφρικής πέρυσι. Πέρυσι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η διεθνή κοινότης κατηγορήθηκε ότι δεν έκανε πολλά πράγματα και ότι έκανε το έκανε αργά. Είδαμε τα μηνύματα στο ΣΑΕΛ τον Νοέμβριο, κινητοποιήσαμε τις πηγές χρηματοδότησης, μέχρι τώρα λειτουργήσαμε έγκαιρα, αλλά δεν είναι επαρκή όλα αυτά. Ξέρετε ότι η έγκαιρη προειδοποίηση απαιτεί δράση, κινητοποιήσαμε 285 εκατομμύρια ευρώ, 350 εκατομμύρια δολάρια δηλαδή, και σε, με συνεργασία με τους Αμερικανούς φίλους μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε και επιπλέον χρηματοδότηση. Αλλά απαιτείται να γίνουν ακόμα περισσότερα. Η πρώιμη δράση στον τομέα αυτό απαραίτητη είναι για να σώσει ζωές αλλά και δεν πρέπει να είναι ε, αποκλειστικά κάτι το ακριβό. Νομίζω ότι η προμήθεια τροφών μπορεί να γίνει με τιμές οι οποίες είναι ε, σχετικά συμφέρουσες. Αν περιμένουμε όμως καιρό τότε τα τρόφιμα γίνονται πιο σπάθια και ακριβένουν και τότε η ανθρωπιστική βοήθεια θα είναι ε, λιγότερο αποτελεσματική γιατί με τα ίδια χρήματα θα αγοράσουμε λιγότερα τρόφιμα. Είναι λοιπόν ε, σωστό να αγοράσουμε τα τρόφιμα σε αποδεκτές τιμές έτσι ώστε να καλύψουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κρίση αυτή που είναι μια κρίση τροφίμων. Γνωρίζουμε ότι το να αντιμετωπίσει κανείς ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει κάποια πρώτα μικρά προβλήματα είναι λιγότερο ε, κοστοβόρο από ότι να καλύψει τις ανάγκες ενός παιδιού που έχει πλέον ασθενήσει από την αδυναμία. Λοιπόν, όλες οι δράσεις μας λοιπόν εντάσσονται σε ανθρωπιστικές ευρωπαϊκές δράσεις, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες που ξέρετε, τρόφιμα, πρόσβαση σε τρόφιμα, ε, κάλυψη τροφιμικών αναγκών από τις τοπικές αγορές κτλ. Αυτό που δημιουργεί προβλήματα είναι η κατάσταση στο Μαλή, στον Ήγυρα ε, και ένας από τους φόβους μας είναι ότι αυτά που συνέβουσαν στο Μαλί ε, κάποιοι από τους εταίρους μας θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα ε, για να βοηθήσουν αυτούς οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί από την κρίση στον βορρά ε, του Μαλί και τη σύγκρουση ανάμεσα στους, στους επαναστάτες και την κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσέθεσε 9 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση της κρίσης των εκτοπισμένων στο Μαλί και να βοηθήσουμε έτσι και τις δυνατότητες των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εκεί. Η κατάσταση όμως εξελίσσεται. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε προβλήματα στα τρόφιμα, ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση στα τρόφιμα, οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται συνεχώς και ε, δεν έχουμε και εύκολη πρόσβαση σε αυτούς που θέλουμε να βοηθήσουμε λόγω της ανασφάλειας. Είναι απαραίτητη λοιπόν η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά δεν είναι ε, ε, η μοναδική. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι βραχυπρόθεσμη ανταπόκριση για να σώσουμε ζωές. Αυτό που απαιτείται όμως είναι να αντιμετωπίσουμε τα βασικά προβλήματα της τροφιμικής κρίσης στην περιοχή που κρατάει πάνω από 10 χρόνια και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας και μέσω της συνεργασίας των κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση του Τσάφ δεν ανταποκρίνεται σωστά για να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών της, το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια μηνύματα θετικά, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε μια μελλοντική νέα κρίση τροφίμων στο ΣΑΕΛ μόνο αν η ασφάλεια ε, πρόσβαση στα τρόφιμα είναι εγγυημένη, αν υπάρξει ουσιαστική αναπτυξιακή βοήθεια για τη γεωργία, έτσι ώστε να παράγει όχι για εξαγωγές μόνο, αλλά για την κάλυψη των τοπικών αναγκών με συνδυασμό μεσοπρόθεσμων και ε, μακροπρόθεσμων μέτρων. Ήταν πολύ καλό το ότι πήγατε και εσείς οι ίδιοι στο Τσάδα, από ό,τι κατάλαβα από την παρουσίασή σας Αυτά τα οποία κάναμε μέχρι τώρα ήταν απαραίτητα αλλά δεν ήταν επαρκή και μένει ακόμα πολλά να γίνουν. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Κόρη της UNICEF. Θα ήθελα, αν θέλετε, να σημάνω μια κρίση ανάγκης να συνειδητοποιήσετε όλοι. Όπως είπατε, Πρόεδρε, εσείς η ίδια, Αποφασίζουμε σήμερα για την καταδίκη ε, άνω του εντός εκατομμυρίου παιδιών που υποφέρουν από την έλλειψη τροφής και τον υποσυτισμό. Το θέμα δεν είναι μόνο ε, κάποια τρόφιμα, ακόμα και αν ε, δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στην ύπαρξη των τροφίμων από τη μία και τον υποσυτισμό από την άλλη. Λοιπόν, σήμα κινδύνου προς όλους ε, τους ε, ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε πάρα πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις τηλεοράσεις μας. Η κοινή γνώμη δεν είναι ενημερωμένη. Απαιτείται δράσεις και αυτό το υπογράμμισε και ο εκπρόσωπος της ΕΚΟ. Έχουν δοθεί τρόφιμα και σχετικά με την αποτελεσματικότητα του κόστους. Αν αν εμείς δώσουμε αυτό το, αυτή την τροφή η οποία βασίζεται σε, παράγεται από φιστίκια, τότε θα γλιτώσουμε ε, κόστος δεκαπλάσιο στο μέλλον για να καλύψουμε τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν. Για μας λοιπόν το θέμα δεν είναι μόνο να σώσουμε τις ζωές των παιδιών, κάτι το οποίο έτσι και πρέπει να κάνουμε, το θέμα είναι να προσπαθήσουμε εμείς να μην χαθεί μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων η οποία χρειάζεται πάρα πολύ. Ακόμα και σε περίοδους κρίσης, πριν από την ηλικία των δύο παιδιών, όταν υπάρχει υποσυτισμός, επηρεάζεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού ανεπανόρθωτα. Επηρεάζεται η ικανότητα του παιδιού να αναπτυχθεί ακόμα και αργότερα, όταν θα έχει ας πούμε τρόφιμα. Λοιπόν, γι' αυτό επιμένουμε στα θέματα της διατροφής. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα βάχη πρόθεσμα και μακρο μακροπρόθεσμα και πρέπει να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν ε, τα παιδιά αυτά σωστά, να είναι ανθεκτικά. Ξέρουμε ότι ένα υποσύτημένο παιδί ε, όταν χάσει και ότι θα χάσει δύο-τρεις χρονιά στο σχολείο. Ξέρουμε ότι οι χώρες που υποφέρουν από υποσυτισμό ή που έχουν υποφέρει από υποσυτισμό ε, θα χάσουν δύο ή τρεις πόντους του ΑΕΠ τους για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του υποσυτισμού. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία γνωρίζουμε πως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν δίκτυα τα οποία πρέπει να κινητοποιηθούν, μπορούμε να τα κινητοποιήσουμε και θα πρέπει οι προσπάθειες που κάνουμε τώρα να εντατικοποιηθούν, να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Για το Τσάδ, για τον Ήγυρα, η κατάσταση εξελίσσεται βέβαια, για το Μαλί. Έχουμε καλύψει το 90% των αναγκών σε σχέση με αυτό, με αυτό το μικρό τρόφιμο που παρασκευάζουμε από ε, φιστίκια εμείς είμαστε θα έλεγε σε επαφή με τα σημεία ανάγκης και έχουμε ακριβώς ε, κινητοποιήσει τα δίκτυα παροχής αυτών των τροφίμων επιβίωσης και στο Μαλί και στον Ήγυρα. Συνεργαζόμαστε με 20 διεθνείς ε, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και 13 ε, μη κυβερνητικούς τοπικούς εταίρους Έχουμε δημιουργήσει, περάσαμε μέσα σε λίγους μήνες από 3.000 σε 4.000 κέντρα υγείας για να αντιμετωπίσουμε τις πιο σοβαρές περιπτώσεις υποσυτισμού. Η δυνατότητα λοιπόν υπάρχει, αλλά θα πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση προς τα άνω και σε επίπεδο ταμείου και σε επίπεδο δράσης. Απαιτείται συγκεκριμένη παρέμβαση λοιπόν και από πλευρά σα. Έχουμε ανάγκη τη βοήθειά σα. Ε, το θέμα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το θέμα είναι να φέρουμε σε επαφή τους σωστούς εταίρους και η συνεργασία μας με την ΕΚΟ είναι καλή. Κάποιες χώρες μέλη και η ΕΚΟ ιδιαίτερα αντέδρασαν γρήγορα και ξέρουμε τι μαθήματα, από τα μαθήματα που πήραμε πέρυσι πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να καλύψουμε μια εξελισσόμενη λοιπόν κατάσταση μπροστά μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας Ελπίζω και εσείς οι λίγοι κοινοβουλευτικοί να προσπαθήσετε να βοηθήσετε στην κινητοποίηση της κοινή γνώμης, της διεθνούς κοινότητας και όσους άλλους μπορούν να βοηθήσουν. Πρόκειται για μια κρίση διατροφής για τα παιδιά. Πρόκειται για μια κρίση που αφορά τη νέα γενιά των παιδιών της Αφρικής, αυτής της περιοχής του Σαέλ. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κορή. Συμφωνώ απόλυτα με όσα μόλις είπατε. Αντίθετα λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να απευθυνθούμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι συντελείται αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή με την ε, ε, κατάσταση αυτή που περιγράψατε ε, του υποσυντισμού των παιδιών. Θα έρθουμε λοιπόν ταχύτατα τις επόμενες μέρες επαφή μαζί σας. Να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου, τον κύριο Κορτές Λάστρα. Κυρία Πρόεδρε, λίγα μπορώ να πω που δεν έχετε ήδη πει. Πήγατε στην Κένια, πήγαμε και στο Κέρας Αφρικής. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αύριο θα έχουμε και την Επίτροπο Γεωργίευα εδώ και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τις προσπάθειες που... Α, όχι! Νόμιζα ότι θα ερχόταν. Ε, αύριο είναι ο δομημένος διάλογος, ε, τέλος πάντων. Αλλά θα αναφέρουμε και αυτό ε, στην κυρία Γιώργη. Δεν θα χαρεί ιδιαίτερα, τέλος πάντων. Ναι, θα τις κάνουμε ερώτηση και για αυτή την κατάσταση, το λιγότερο. Λοιπόν, Πράγματι γίνονται σημαντικές προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταβάλουμε προσπάθειες, προσπαθούμε να πετύχουμε ό,τι μπορούμε. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν κατάλαβα καλά ποια είναι η κατάσταση της διεθνούς συντονισμένης ανταπόκρισης. Είπατε ότι υπήρξε ένα συνέδριο. Προβλέπονται και άλλα συνέδρια για το μέλλον. Η σχέση και ο συντονισμός με Τη είπα τι γίνεται, γιατί αν ε, μάλλον με, τις, ε, με τα Ηνωμένα Έθνη ε, υπάρχει, ακούμε και διαβάζουμε Γιατί τη Μαυριτανία, για το μάλλον για άλλες χώρες. Αλλά συντονισμός υπάρχει για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά και πιο συντονισμένα σε τέτοιες ε, καταστάσεις που ανακύπτουν συνεχώς και που έχουν πραγματικά τεράστια σημασία τουλάχιστον για την Επιτροπή μας και για τους βουλευτές που την απαρτίζουν. Αυτή είναι η ερώτηση προς την Κομισιό. Σας αφήνω να απαντήσετε, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Είναι πάρα πολύ ευστόχο. Είχαμε και εμείς κάποιες ανησυχίες για το συντονισμό. Πράγματι, από την αρχή ε, είδαμε ότι λείπει αυτός ο πραγματικός συντονισμός και πιέσαμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να υπάρξει συντονισμό μεταξύ Ηνωμένων Εθνών, Διεθνών Οργανισμών ε, και Δωρητών, Χρηματοδοτών. Αρχές Φεβρουαρίου, ω Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητήσαμε να γίνει αυτή η συνδιάσκεψη, αυτό το συνέδριο, για να δείξουμε ότι σε διεθνέ επίπεδο κανένα άλλο δεν παίρνει πρωτοβουλίε. Θα περίμενε κανεί ε, και η Ότσα και τα Ηνωμένα Έθνα να αναλάβουν την πρωτοβουλία. Αλλά η Επίτροπο Γεωργίευα είναι αυτή η οποία έγραψε και στην Ότσα και στο UNDP για να αναλάβουν το συντονισμό αυτό, κάτι που έχει γίνει. Πλέον υπάρχει ένας περιφερειακός συντονιστής που προσπαθεί να συντονίσει εθνικές πρωτοβουλίες και άλλη ε, προσπάθεια ήταν να συνδέσουμε την βράχη πρόθεσμη με την, ε, μακρο, με την ε, μακροπρόθεσμη. ΟΤΣΑ δηλαδή και UNDP. Δεύτερο σκέλο είναι οι δύο προσεγγίσει, βράχη πρόθεσμη, μάκρο με να συντονιστούν και να συνδυαστούν. Έχουμε λοιπόν ήδη σημειώσει πρόοδο. Θα ήταν όμω πρόημο να πούμε ότι η πρόοδο αυτή μα βοηθά να λύσουμε τα προβλήματα. Είμαστε απλά στη σωστή κατεύθυνση, στο σωστό δρόμο, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Εγώ από πλευρά μου δεν θα πρόβω σε κάποια συμπεράσματα. Πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να γίνουν ε, ορισμένα πράγματα γιατί υπάρχει το ανθρωπιστικό σκέλος. Αυτή η κρίση, η καταστροφή. Πήγαμε στη Γένεια, στη Βόρεια Κένια, αλλά αυτό που είδαμε στο Τσάντα υπερβαίνει κατά πολύ οτιδήποτε έχω δει μέχρι τώρα όσο καιρό είμαι εισηγήτρια για ανθρωπιστικά θέματα. Ήταν πραγματικά φρικτά αυτά που είδαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο μας έχει απομείνει. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τη μερισιά διάταξη. Άρα, ναι. Όχι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Θα διακόψουμε και θα παραλάβουμε αύριο στην ίδια αίθουσα στις 9 ακριβώ στη συνεδρίασή μα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.